Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε. Καθίστε παρακαλώ. Uh, Μία ανακοίνωση έχω μόνο του Προέδρου. Το σημείο 7, τελευταία στιγμή, ζητήθηκε από τη Ρουμανική τηλεόραση να ε, μαγνητοσκοπηθεί η συνεδρίασή μας. Τι λένε οι συνήθεις κανόνες. Είναι δημόσια συνεδρίαση και βγαίνει στο διαδίκτυο. Οπότε δεν μπορεί κανείς να προβάλλει ε, αντίρρηση αφού είναι δημόσια συνεδρίαση. Απλώ σας λέγω ότι θα τραβήξουν ε, κάποια πλάνα από τη ρουμανική τηλεόραση, αλλά έτσι και αλλιώ βγαίνει στο διαδίκτυο. Πάμε στο σημείο 7. Έχουμε μία ώρα για τη συζήτηση. Ανταλλαγή απόψεων Συνάδελφοι. Ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση λοιπόν στη Ρουμανία. Στην Ολομέλεια στις 8 Ιουνίου ζητήθηκε και στις 11 Ιουνίου στη διάσκεψη των Προέδρων. Στόχος είναι να ανταλλάξουμε απόψεις με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς ενώπιόν μας. Πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς ε, έχει έρθει για να ανταλλάξουμε απόψεις. Μας ζήτησε ο πρόεδρος Σούλτς από την Επιτροπή μας να συζητήσουμε ε, για ε, την διεύθυνση καταπολέμησης της διαφθοράς στη Ρουμανία που έχει κινήσει ε, μια έρευνα κατά του προέδρου του, της κυβέρνησης Βίκτορ Πόντα. Στις 8 Ιουνίου λοιπόν το αίτημα αυτό διαβεβάστηκε στην Ολομέλεια και στη συνέχεια στις 11 του μηνός η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή μας για ανταλλαγή απόψεων. Ε, προσκάλεσα τον πρώτο αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων και δέχτηκε αμέσως την πρόσκληση αυτή. Ε, ήταν η πρώτη ευκαιρία που μπορούσε να έρθει και χάρηκα πάρα πολύ που απεδέχθη την πρόσκληση. Έχετε το λόγο κύριε Τίμερμανς και οργανωτικά συνάδελφοι θα ήθελα να σας πω ότι θα δώσω το λόγο αμέσως μετά στους συντονιστές και αν επιτρέψει ο χρόνος στα υπόλοιπα μέλη που θα επιθυμήσουν να μιλήσουν. Φράνς, έχεις το λόγο και ευχαριστώ που ήρθατε. Thank you very much um, for your invitation and um, Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Εφόσον με καλέσατε, ευχαρίστως ήρθα για να καταθέσω για την κατάσταση στη Ρουμανία και μάλιστα βρισκόμουν εκεί πριν από 15 μέρες, την ίδια μέρα μάλιστα, που ο Πρωθυπουργό Πόντα ενημερώθηκε από τις δικαστικές αρχές ότι θα γινόταν ε, έρευνα για τον ίδιο και φυσικά η πρώτη παρατήρηση, όπως καταλαβαίνετε, το είπα ήδη όταν ήμουν στη Ρουμανία γιατί έλαβα πολλά ερωτήματα, η Κομισιόν φυσικά δεν προφανώς δεν είναι σε θέση να σχολιάζει με μονομένες υποθέσεις, αλλά ούτε και να μπει μέσα στις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Αυτό που θέλουμε είναι η δικαιοσύνη να μπορέσει να εργαστεί ανεξάρτητα Από ό,τι φαίνεται η δικαιοσύνη μπορεί να ενεργήσει και να δράσει σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης στη Ρουμανία και όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος ήδη γράψαμε στην τελευταία μας έκθεση σχετικά με την Ρουμανία ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες ενίσχυσης του κράτους δικαίου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο, ε, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι βιώσιμο, αν έχουν φτάσει στο σημείο που δεν υπάρχει γυρισμός ή όχι. Ε, ε, και γι' αυτό θα είμαστε σαφείς, το είπα και δημόσια, το είπα σε όλους τους πολιτικούς που συνάντησα στο εκτελεστικό και στο κοινοβούλιο ότι η Κομισιόν πολύ συγκεκριμένα θα παρακολουθήσει τον ε, διαχωρισμό των εξουσιών στη Ρουμανία και θα μεριμνεί ώστε οποιαδήποτε ενέργεια κάνει το Κοινοβούλιο να μην επηρεάζει την ελευθερία κινήσεως του δικαστικού σώματος και της δικαιοσύνης. Βεβαίως τα διάφορα τμήματα της κυβέρνησης έχουν φέρνει τις ευθύνες τους ε, και αφού μίλησα στους ε, ε, προέδρους των σωμάτων της, της, της Ρουμανίας ε, είπα ότι θα αναλύσουμε τις τροπολογίες ε, για να δούμε κατά πόσο αυτές περιορίζουν τις εξουσίες του, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και από τις επιστολές που έστειλα και από τις ε, συζητήσεις με τους δύο προέδρους, κάποιες από τις ε, τροπολογίες είναι υποσυζήτηση, δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ψηφοφορία. Θα παρακολουθήσουμε πολύ πολύ προσεκτικά το ότι ε, αναφέρεται και στο να μην υπάρξει καμία επίθεση εναντίον του δικαστικού σώματος. Μίλησα επίσης στα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά και σε μια δημόσια συζήτηση που είχα για τη, ε, στα σύνορα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη για τον μηχανισμό CVM, τον μηχανισμό συνεργασία και επαλήθευσης για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και ότι ε, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο στο πλήρες του, στην πλήρη του ισχύ και δυναμικό, γιατί έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αξιοσημείωτη, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κατάλληλο σημείο στο να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Πιστεύω ότι οι αρχές της δημόσιας διαβούλευσης και του σεβασμού στον ρόλο αλλήλων ε, και η πρόθεση όλων αυτών από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα βοηθήσουν τη Ρουμανία να καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση και μετάβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω πρώτα το λόγο σε όποιον εκ των συντονιστών επιθυμεί να λάβει τον λόγο η ε, κυρία Χολμάιρ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρώτα, απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προφορίες που μας έδωσε η ανησυχία που επιθυμώ να εκφράσω σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Ρουμανία προέρχεται από ειδήσει, κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, που λένε ότι προάγονται κάποια νομοσχέδια στην Ρουμανία τα οποία στηρίζουν την διαφθορά και επιτρέπουν διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων για το μέλλον. Για μένα έχει και για σημασία κάτι τέτοιο και για την Ουγγαρία και για την Ρουμανία. Δεν με ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτά τα πράγματα ε, για το ποια πρόσωπα εμπλέκονται θα τα ξεκαθαρίσει η ίδια η Ρουμανία. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή και συμπεριφορές που ενδέχεται να οδηγήσουν στο ενδεχόμενο στη Ρουμανία να επανεμφανιστούν φαινόμενα διαφθοράς συγκρούσεων συμφερόντων που θα αντιτίθεται στα κριτήρια της Κοπενχάγης και στα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση που στην οποία καταλήγω μετά από τις ειδήσει των τύπων αλλά και από πληροφορίες που μου διαθέτουν συνάδελφοι, είναι με την μη άρση της ασυλίας επηρεάζεται η δυνατότητα της δικαιοσύνης. Να μπορέσει δηλαδή να διεξαγάγει έρευνες εναντίον ουδήποτε. Ποιες δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτρέψει τέτοια συμπεριφορά ακόμα δηλαδή και αν γίνεται μέσα σε κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ένα. Έχετε εξάλλου γνώση εάν με νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνε να άρουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που με απασχολούν. Λέω καθαρά εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι τίτλοι των εφημερίδων. Μας ενδιαφέρει να ρηχτεί φως σε οποιαδήποτε υπόθεση. Επαναλαμβάνω τα ίδια που έχουμε πει και για την Ουγγαρία. Θέλω να υπάρξει μια διαρκής στήριξη μιας τακτικής και τακτοποιημένης δικαιοσύνης και των ποινικών διαδικασιών, μιας διαδικασίας βασισμένης στις δημοκρατικές αρχές που να εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να μην τις προβάλλει κολλήματα. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα για μένα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Βίργκιτ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ και εγώ. Πρώτα θα συμφωνήσω με την κυρία Χόλμαϊερ ότι δηλαδή όταν πρόκειται για υποθέσεις διαφθοράς ή για άλλα ατοπήματα ακόμα και αν αυτά βαρύνουν πολιτικούς καταρχήν είναι θέματα τα οποία πρέπει να επιλύονται στο εθνικό επίπεδο. Στο παρελθόν είχαμε υποθέσεις όχι μόνο στην Ουγγαρία και Ρουμανία, αλλά και σε πολλές από τις λεγόμενες παλαιές χώρες μέλη, στη βάση των οποίων είχαμε μάλιστα ασκήσει κριτική. Το ερώτημα που τίθεται για μας τώρα είναι υπάρχει διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά πράγματα και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω λοιπόν μια ουσιαστική ερώτηση για τον Φρανς Τίμερμανς, εάν μπορεί να την απαντήσει, διότι όσον αφορά την υπόθεση Πόντα, ακούγονται διάφορες μομφές και επίκαιρες αλλά και κάποιες που ανάγονται σε παρελθόντα έτη. Αν οι προφορίες μου είναι σωστές, στις περιπτώσεις που ανάγονται στο 2007 διεξάγονται όντως έρευνες ανεξαρτήτως της άρσεως της ασυλίας. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι λειτουργεί το σύστημα της δικαιοσύνης. Τώρα με ποια αιτιολογία δεν ήρε την ασυλία η Ρουμανική Βουλή, νομίζω ότι αυτό εκφεύγει την αρμοδιότητα μας γιατί είναι θέμα της Εθνικής τους Βουλής. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και που άπτεται του ποινικού δικαίου είναι ουσιώδους τύπου. Εφόσον κάποιος αξιωματούχος συμπεριφέρεται εσφαλμένα, ενδεχομένως μάλιστα δωροδοκείται. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θυμάμαι, είχαμε σχετικές εκθέσεις για τις περιπτώσεις διαφθοράς βουλευτών ή και υπουργών. Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα στάνταρ είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Θα έπρεπε να τα εξετάσουμε για να μπορούμε να προβούμε σε μια σύγκριση και θα πρέπει να δούμε υπάρχουν πράγματα τα οποία όντως φύγουν το ευρωπαϊκό δίκαιο ή οφείλουμε να επαφεθούμε στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χώρες μέλη. Ελπίζω η σημερινή συζήτηση να διευκολύνει την απάντηση ορισμένων ερωτημάτων. Ταυτόχρονα η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι σε θέματα κράτους δικαίου και σε θέματα τηρήσεως ορισμένων βασικών αρχών όντως υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης σε πολλές χώρες μέλη και σε πολλούς τομείς και στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να διακρίνουμε με μονομένες περιπτώσεις από περιπτώσεις που έχουν διαρθωτικό χαρακτήρα και με ποια διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συντονιστές εγγεγραμμένους. Δείξτε μου, εάν θέλετε να λάβετε το λόγο, Άννα Γκόμης, Μακιαβέλη, Σόε. Καλά, καλά. Σιγά σιγά. Ένας, ένας λοιπόν ή μία μία. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Θα επανέλθω μετά. Ο κ. Κουέλιο δεν ε, επιθυμεί να μιλήσει. Ωραία. Συλλέγει τα ονόματα ο πρόεδρος. Sorry. Um, Άλλος κανείς από την πλευρά αυτή. Ας πάρουμε τώρα με τη σειρά. Η κυρία Μακοβέη. Η Άννα ήταν πρώτη. Ωραία, Άννα, εσύ ζητήσατε πρώτη το λόγο. Ωραία, αρχίστε. Δεν γνωρίζω τα της υποθέσεως, τι συνέβη στη Ρουμανία μόλις άκουσα τις πληροφορίες του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ανησυχεί που βλέπω ότι διεξάγονται έρευνες και ταυτόχρονα προσπάθειες να τροποποιηθούν οι διαδικασίες με τρόπο που όντως θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη οι και να υπονομευθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης. Προέρχομαι από μια χώρα, εννοεί την Πορτογαλία, όπου ο πρώην ηγέτης του κόμματο μου και πρώην Πρωθυπουργό είναι στη φυλακή. Ήποπτο για διαφθορά. Η γραμμή που πήρε το κόμμα μου ήταν αυτή τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Και θα ήταν απολύτω αδιανόητο να προαχθούν οποιασδήποτε αλλαγέ για να αλλάξει το σύστημα τη δικαιοσύνη που ασκεί ε, διώξεις και δεξαγέρευε. Θα ήταν απολύτω απαράδεκτο κάτι τέτοιο. εφόσον είναι απαράδεκτο στη χώρα μου, βεβαίω θα πρέπει να είναι απαράδεκτο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλο τη Ένωση. Ελπίζω και εύχομαι η Κομισιόν να παίξει σημαντικό ρόλο. Ομολογώ ότι η προηγούμενη Επιτροπή, η προηγούμενη Κομισιόν δηλαδή, μα είχε απογοητεύσει σε θέματα διαφθορά. Εγώ είχα θέσει ορισμένα θέματα διαφθορά με υψηλέ ευθύνε και στην ίδια Επιτροπή και στον ίδιο τον κύριο Μπαρόσο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έπραξε τίποτε. Μέχρι σημείου που η συνήγορος του πολίτου πρόσφατα επέστρεψε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντηση μάλλον, ρωτώντας πώς είναι δυνατόν να μου δίνει τέτοιες απαντήσεις σε ερώτησή μου. Και αναφέρονταν σε υποβρύχια που είχε αγοράσει ο ε, πρόεδρος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν τότε υπουργό Άμυνα, και αυτά οδήγησαν σε καταδίκες στη Γερμανία ενώ στην Πορτογαλία ακόμα δεν έχουν βρεθεί ε, τα διεφθαρμένα πρόσωπα. Αυτό ήταν το παράπονο μου, αυτή ήταν η καταγγελία μου δηλαδή και μετά οι καταγγελίε που έκανα για την επαναδιαπραγμάτευση των λεγόμενων offset, των παράπλευρων ωφελών δηλαδή και ούτω καθεξή. Δεν εδόθηκε καμία συνέχεια σε αυτά τα πράγματα. Και μόνο μια μικρή υποσημείωση στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ είχα άξορα εκ των υστέρων ότι πρόκειτο για ε, προβλεπόταν ολόκληρη σελίδα. Ε, θα ρωτήσω λοιπόν κύριε Αντιπρόεδρε, να παρακαλέσω μάλλον κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμερμανς. Παίξτε τον όλο σας. Ε, φανείτε σκληρός. Να μάλιστα σκληρός, λέει ο πρόεδρος. Εγώ μπορώ να μην σου αλλά για πολύ λίγο. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά η καθεμία ή ο καθένας. Λοιπόν, δύο λεπτά ο κάθε συνάδελφος και η κάθε συνάδελφος και ακολουθεί η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Περιμένω και εγώ απάντηση ε, σε ένα mail που σας είχα στείλει και θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας το εξής. Η Ρουμανία ήδη ε, έχει πληγεί πολύ ως προς το κύρος, το γόητρο και την εικόνα της. Το ξέρει και ο πληθυσμός της χώρας ότι ο Πρωθυπουργό διώκεται, είναι σε επίσκεψη στην Τουρκία σήμερα και κάποιος του είπε ότι δεν δικαιούται να παραμένει Πρωθυπουργό. Και οι ίδιοι οι Ρουμάνοι κάπως έχουν ενοχληθεί από το γεγονός ότι επικαλείται την ασυλία του και παραμένει πρωθυπουργός. και ε, η δικαιοσύνη ε, και ο ποινικό ε, κώδικας θα πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορούν να γίνονται αλλαγές έτσι, στα γρήγορα με στόχο να παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης. Επίσης είπατε ότι αξιολογείται τη Ρουμανία διότι αυτός ο μηχανισμός είναι στις δικές σας αρμοδιότητες. Ο μηχανισμός για τη ε, συνεργασία και την επαλήθευση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια τα ίδια. Ότι οι θεσμοί ε, κάνουν τη δουλειά τους, οι δικαστές και οι εισαγγελείς εννοώ, η δικαιοσύνη στη χώρα, αλλά τι γίνεται με την πολιτική βούληση να παταχθεί η διαφθορά. Εκεί είναι το πρόβλημα δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την ε, συμπολίτευση, από την πλειοψηφία. Αυτό από το 2012. Κοιτάξτε όλες τις εκθέσεις. 2012, 2013, 2014, 2015 όλα τα ίδια λένε. Από τότε που ε, ήρθε στην εξουσία ο συνασπισμός της οποίας ηγεί το Βίκτορ Πόντα δεν υπάρχει παραμικρή πολιτική βούληση. Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν. Ως προς τη λειτουργία των θεσμών τώρα, δεν γυρίζει πίσω αυτή. Γιατί το λέω. Γιατί μας λέτε ότι δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ επικαλούμε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2012 συγγνώμη, μέχρι σήμερα. Από την άλλη, το Κοινοβούλιο αρνείται να άρει την ασυλία του Πρωθυπουργού και όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για φίλους του ε, του ε, Ρουμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Υπάρχει όμως πρόβλημα με αυτά τα νομοσχέδια ε, και σε ό,τι αφορά για την άρση της ασυλίας είπαμε και ακούστηκε ότι πρόκειται για εθνικό ζήτημα. Να σας αναφέρω και άλλη μία περίπτωση που άπτεται αυτού του μηχανισμού. λέμε και ακούγεται μάλλον ότι θα πρέπει οι πιο ακέραιοι να είναι μέλη της κυβέρνησης. Και δεν μπορούν οι υπουργοί, πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργό, να είναι υπό έρευνα. Οι πιο ακέραιοι λοιπόν χαρακτήρες λέτε και το λέει και η έκθεση του μηχανισμού για τη συνεργασία και την επαλήθευση ε, της Ρουμανίας. Εδώ όμως έχουμε πρόβλημα, διότι αν θέλουμε να είναι οι πιο αδαμάντινοι χαρακτήρες στην κυβέρνηση, πώς θα είναι αφού δεν μπορούμε να άρουμε την ασυλία εκείνων που από ό,τι φαίνεται δεν είναι και παραμένουν. Οι 23 νομοσχέδια λέτε ότι τα έχετε σταματήσει. Και εδώ επικαλούμε ακόμα τα κριτήρια της Κοπενχάγης εδώ. Ε, ήταν 23 νομοσχέδια με στόχο να αλλάξει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο ποινικό κώδικας. Ε, μετά από λίγα χρόνια λοιπόν εφαρμογής ε, αυτών υπάρχουν προβλήματα και εσείς λέτε ότι πρέπει να αλλάξουν και ξαφνικά έρχονται πρωτοβουλίες όλες από την κυβέρνηση και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τα άλλα κόμματα ε, που είναι κυβερνητικό κυβερνητικός συνασπισμός έχουν φέρει ε, νομοσχέδια για να σταματήσουν οι έρευνες. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ο Πρόεδρος, μια στιγμή, να δώσω τα παραδείγματα και θα σταματήσω. Ναι, μια στιγμή. Αν μιλήσετε περισσότερο, δεν θα μιλήσουν οι συνάδελφοί σας. Και είναι θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Γιατί Τώρα έχουμε 7 ή 8 συναδέλφους από την ίδια σα την ομάδα. Αν συνεχίσετε εσεί, τελειώνω, τελειώνω. Έλεγα λοιπόν 23 νομοσχέδια προσπαθούν να σταματήσουν αυτή την προσπάθεια. Μεταξύ άλλων προβλέπουν να μειωθεί σημαντικά η δυνατότητα ε, παρέμβασης για αυτόφορο. Γίνεται μια εξάμηνη ε, ρύθμιση, προθεσμία για να ε, γίνονται οι καταγγελίες για δωροδοκία γιατί 6-8 μήνες και μετά δηλαδή θα παραγράφονται. Ε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εάν ένας εισαγγελέα ε, θεωρήσει ότι υπάρχει κατάχρηση εξουσίας κινδυνεύει να διωχθεί. Επαναλαμβάνω, 23 νομοσχέδια προσπαθούν να επέμβουν στη δικαιοσύνη. Μέσα Ιουλίου είναι η καταληκτική προθεσμία. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Αν δεν τους δώσω το λόγο θα προσβληθούν οι συνάδελφοι, θα στεναχωρηθούν. Ε, γι' αυτό ανησυχώ. Κανένας δεν θα πρέπει να θεωρείται ε, αδικημένος. Παρακαλώ να τηρείτε το δίλεπτο συνάδελφοι και αν έχουμε την ευκαιρία θα ξαναμιλήσετε. Ε, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμας, μίλησε λιγότερο από όλους. Ε, αν έχουμε χρόνο θα ξαναμιλήσετε. Ο Βίκτορ Μποστινάρου είναι επόμενος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να μιλήσω ρουμανικά και να αναφερθώ πρώτον την πάρα πολύ ισορροπημένη σας και αντικειμενική κρίση, όσο και ουδέτερη ε, στα σχόλιά της για την κατάσταση στη χώρα μου. Θα μιλήσω λοιπόν ρουμανικά. Πρώτον, λυπάμαι πάρα πολύ που άλλη μία σύγκρουση ρουμανο-ρουμανική εκτελήσεται στην Επιτροπή Ελευθεριών ε, και μάλιστα με τα ίδια πρόσωπα και ε, ε, πρωτοβουλία του ίδιου προσώπου. Και το πρόσωπο που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση έχει μάλλον αμφισβητούμενη πολιτική νομιμότητα, αφού έλεγε ότι έγινε νοθεία 1,5 εκατομμυρίων ψήφων στο δημοψήφισμα. Και τώρα γίνεται λόγος για 70 άτομα. 70 άτομα που ενδεχομένως να ε, ε, μην ψήφισαν όσο όφυλαν. Για το 2006, 2007, 2008 πρόκειται αυτή η περίπτωση ε, για τον Πρωθυπουργό που το 2012 κατέληξε υπό την ένδοξη προεδρία του Τραϊάν Μπασέσκου. Και ελήφθη η απόφαση να μην αρθεί η ασυλία του. Εγώ δεν θέλω να σχολιάζω ε, αποφάσεις κοινοβουλίων, ακόμα και αν είναι το κοινοβούλιο της ίδιας μου της χώρας. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν σχέδια τροποποίησης της νομοθεσίας ε, στη Ρουμανία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται ε, να αξιολογήσει αν είναι σωστές οι προτάσεις αυτές για τις καταχρήσεις και για τις κυρώσεις ε, που θα επιβάλλονται σε όποιους ε, παραβαίνουν. Δηλαδή όταν κάποιος παυθεί για 6,5 μήνες ας πούμε και δικαιωθεί ε, και αθωωθεί από την απόφαση, τι γίνεται στη συνέχεια. Επίσης η τροποποίηση της νομοθεσίας ε, θέλει να τερματιστεί αυτό το θέαμα ε, των ανθρώπων με χειροπέδες που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ξέρω ότι στη χώρα σας κύριε Τίμερμανς, στη Γαλλία, στη Σουηδία, όλα αυτά εκδικάζονται στα δικαστήρια και όχι στην τηλεόραση. Μία από τις προτάσεις λοιπόν φιλοδοξεί να σταματήσει αυτό το θέαμα, αυτή η περιφορά, αυτό το, το ενοχλητικό και άχαρο θέαμα των ανθρώπων με χειροπέδες να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Αυτό είναι θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης, θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει την ίση μεταχείριση και να έχουν την ίδια μοίρα και οι... όσοι δωροδοκούν και όσοι δωροδοκούνται, όσοι χρηματίζουν και όσοι χρηματίζονται. Το είπε και η κυρία Γκόμες. Στη Ρουμανία δεν έχουμε ισότιμη μεταχείριση των δύο πλευρών, γιατί στη διαφορά χρειάζονται δύο. Και δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία αυτό. Θα πρέπει να ληφθεί μια δέσμη μέτρων για όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει ένα phasing out για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και να γίνεται σωστά η τήρηση των νόμων παντού. Yeah, thank you, Chair, and uh, thank you, Commissioner, for attending. Uh, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ, ε, Πίτροπε, που είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Με εξέπληξε κάπως το ότι άκουσα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα εθνικό θέμα. Είμαστε έτοιμοι να αναμειχθούμε σε έναν πόλεμο, έναν ε, πόλεμο πολιτικό στη Ρουμανία. Διερωτώ με από πότε το να προσπαθεί κανείς να εμποδίσει τη δικαιοσύνη είναι εθνικό θέμα. Μάλιστα πρόκειται για νομικό ζήτημα και πολύ σοβαρό, γιατί το να χρησιμοποιεί κανεί δημοκρατικά μέσα για να περιορίσει στην ουσία τη δημοκρατία δεν είναι εθνικό θέμα, είναι ένα πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα. Για να δουλέψει η δημοκρατία εναντίον του εαυτού τη μέσω μια κοινοβουλευτική ψηφοφορία πάλι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί όχι μόνο είναι διεφθαρμένο, αλλά είναι και επικίνδυνο και σίγουρα δεν είναι ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και είναι σωστό το ότι γίνεται η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ Μέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ την ευκαιρία για να σας μιλήσω στα ουγγρικά, γιατί έτσι θα είναι και περιπέτεια για σας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν κατάλαβα ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Από ό,τι άκουσα, το Ρουμανικό Κοινοβούλιο δεν έχει αποσύρει την ασυλία του Πρωθυπουργού. Το Ρουμανικό Κοινοβούλιο γνωρίζει μάλλον γιατί δεν την είδε την ασυλία. Και δεν κατάλαβα γιατί εμείς εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε αν ναι ή όχι θα πρέπει να έρθει την ασυλία του Πρωθυπουργού το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στη διερμηνία. Όχι, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω το λόγο ή με αφήνετε να κλείσω. Όχι, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην διερμηνία. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ακούσαμε επίσης ότι υπάρχουν και διάφορα νομοσχέδια. Νομοσχέδια τα οποία μελετά το Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές, διότι ε, πρόκειται για... είναι μάλλον νομοσχέδια που είναι υποσυζήτηση και έπειτα. Ακούω εδώ και μέρες γιατί πρέπει εμεί να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των χωρών. Γιατί να μην αφήσουμε το Κοινοβούλιο να ρυθμίσει τα προβλήματα αυτά. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο νομίζουμε εμείς εδώ ότι είναι το δικό μας καθήκον. Από τη μια πλευρά άκουσα ότι υπάρχει μια έντονη διαστηριότητα κατά τη διαφθορά από το δικαστικό σώμα της Ρουμανίας. Πολλοί έχουν συλληφθεί, άρα το δικαστικό ε, σώμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί. Γιατί λοιπόν εμείς εδώ πρέπει να το συζητάμε. Εγώ πιστεύω θα έπρεπε, και η κυρία Χολμάγερ το είπε ότι διάβασε στις εφημερίδες το τι συμβαίνει, ίσως θα έπρεπε λοιπόν να εμβαθύνουμε στα ζητήματα για να δούμε ποια είναι, ποια είναι ε, τα αδικήματα περί των οποίων πρόκειται. Αν ας πούμε έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, ε, οι δικαιώματα. Εφόσον δεν ισχύει κάτι τέτοιο και συνεχίζεται η δικαστική έρευνα, θα έλεγα ότι εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο Σόγκορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ζω στη Ρουμανία, πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Αν σκεφτώ τώρα ότι ο ενεργεία πρωθυπουργός είναι πρώην στρατηγός και ότι ο μελλοντικό αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ίσως να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, Ξέρουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στη Ρουμανία άνευ προηγουμένου αποτελέσματα στην καταπολέμηση διαφθοράς. Παρά αυτά τα θετικά αποτελέσματα, οι ετοιμιγορίες, οι αποφάσεις είναι πολύ συχνά ασυνεπείς και πολύ συχνά έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Η δημόσια δίκηση δε της χώρας είναι συχνώς, σχεδόν παραλυμένη γίνονται ε, πολιτικές ε, ενέργειες στο όνομα της καταπολέμησης της διαφθοράς Έπειτα, για να έχουμε μια γενική ιδέα για το τι συμβαίνει στη Ρουμανία, χωρίς να πιέζουμε την Κομισιόν να ερευνήσει για το τι γίνεται εκεί, όπως στην περίπτωση της Ουγγαρίας, Τέταρτον, πολύ ενδιαφέρον ότι το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων πρόσφατα συνέταξε ένα σχέδιο για την ε, ε, στρατηγική δημόσιας ασφάλειας και είπε ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο υπάρχει ε, ότι οποιοδήποτε είδος διαφθοράς είναι απειλή στη δημόσια τάξη. Αυτά, αυτά θέλω να σας, ήθελα να σας τα πω για να έχετε μια γενική εντύπωση για το τι συμβαίνει στη Ρωμανία. Εσύ με το πρωί δεν ζήτησα το λόγο από το ε, ΦΡΑ, δηλαδή τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, γιατί ξέρω τι απάντηση θα μου δώσει. Πάντως, όταν μέλη εθνικών μειονοτήτων ε, ή έχουν προβλήματα ή τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά, παρεμβαίνουν. Αλλά αυτή είναι η απογευματινή συζήτηση, θα επανέλθω ίσως αυτό. Thank you very much. I'll be very short and I will speak. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Θα μιλήσω στα ρουμανικά. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα των κυρίων Μακοβέη και Ουράνου. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι μια βουλή δεν επιτρέπεται να εμποδίζει έρευνες έστω και σε βάρος ενός υψηλού αξιωματούχου διότι αυτές εξυπηρετούν την δικαιοσύνη. Η κατάσταση στη Ρουμανία είναι εξαιρετικά δυσχερής. η πλειοψηφία στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να ανοίξει τον δρόμο στη δικαιοσύνη. Άκουσα σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όλε τις πολιτικές ομάδες ότι νομοσχέδια που αναφέρονται στην ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της ε, δικαιοσύνης που εμποδίζουν την εξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης είναι απολύτως απαράδεκτα. Θα οδηγηθούμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη Ρωμανία. Ούτω ή άλλω υφιστάμεθα πολύ προσεκτικό monitoring, παρακολούθηση δηλαδή και για θέματα δικαιοσύνη. Η κυρία Ρούνατσεκ έχει ζητήσει το λόγο, αλλά ε, δυστυχώ είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων και ε, έχω δώσει το λόγο ή ε, Μαρθά θα λόγο. Κύριος Βοσιτσόφσκι, Βοσιτσιχόφσκι, συγγνώμη, κύριε πρόεδρε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αφού μιλούμε για ρουμανικά θέματα, εγώ δηλαδή αρχικά ήθελα να μιλήσω ως εκπρόσωπος της διακομματικής ομάδας για την προστασία των ζώων, ήθελα να θέσω το θέμα της αντιμετωπίσης, των, της μάλλον, των ζώων στη Ρουμανία, των σκυλιών ιδιαίτερα. Εγώ έχω προβεί σε διαβήματα στην ε, ρουμανική κυβέρνηση, διότι με βάρβαρο τρόπο θανατώνει θα τα ζώα αυτά. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αγανάκτηση και θλίψη του ανθρώπου σε όλη την Ευρώπη και του Ρωμάνους βεβαίως. Αυτό είναι πολύ άσχημο σημάδι για την δράση τη ε, ρουμανικής κυβέρνησης και παρακαλώ να ασκηθούν πιέσεις ώστε να υιοθετήσει πιο φιλόζωες μεταχείρισεις. Ε, ακούω από πολλούς Ρουμάνους ότι και στην υπόθεση αυτή της εξολόθρευσης δηλαδή των αδέσποτων σκυλιών παίζουν ρόλο υποθέσεις διαφθοράς. Φαίνεται ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται διότι για κάθε θανατούμενο σκύλο εισπράττονται αμοιβέ. Μέχρι και 100 και 200 ευρώ από ό,τι φαίνεται. Πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να μας απασχολήσει όλους η Ρωμανία υφίσταται βλάβη στο κύρος της εντελώς περιττή με τον τρόπο αυτό. Οφείλει και αυτό να λυθεί υπόψη, διότι την ευθύνη την φέρουν εδώ οι ρωμανικές αρχές. Διότι ακολουθεί πρακτικές που είναι απολύτως απαράδεξες για τη σημερινή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, λέει ο Έχουν ζητήσει να δευτερολογήσουν οι δύο συντονίστριες, η κυρία Ζίμπλ των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και η κυρία Μάιερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η Μπίργκιτ. Θα είμαι σύντομη. Υπάρχει διαφθορά στην Ευρώπη, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει διαφθορά στη Ρουμανία, επίσης η απάντηση είναι ναι. Θα μπορούσα λοιπόν να συμφωνήσω με τη συνάδελφο ότι η Ρουμανία δείχνει μια σχημή εικόνα. Υπάρχει όμως και ένα καλό μήνυμα. Στην Ρουμανία δηλαδή διεξάγονται έρευνες Εκτός από την υπόθεση Πόντα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κατά των οποίων διεξάγονται έρευνες και πολλοί πολιτικοί μεταξύ αυτών. Αυτό είναι δείγμα του ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε έκθεση επί της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που ακόμα τελούν υπό παρακολούθηση και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βεβαίωσε ότι η Ρουμανία σημειώνει σημαντικά βήματα πρόοδα. Μην το λησμονούμε. Υπενθυμίζω επίση ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε και διαπραγματευόμαστε μια οδηγία για την θέσπιση του τεκμηρίου αθότητα. Αν λοιπόν υπάρχουν υπόνοιε, πρέπει να γίνουν έρευνε. Σωστό. Μέχρι την απόδειξη όμω τη ενοχή, πα άνθρωπο είναι αθώο. Το τονίζω αυτό διότι κάπως αλλιώ τα είπαν ορισμένοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νομοσχέδια που προωθούνται, ναι, πρόκειται για μια ατυχή χρονική σύμπτωση, τουλάχιστον αυτό μπορεί να το πει κανείς. Και εδώ όμως πρέπει να ελεγχθεί με αντικειμενικότητα αν όντως τα νομοσχέδια αυτά οδηγούν σε περιορισμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ναι ή όχι. Εάν συμβαίνει αυτό πράγματι είναι θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά ούτε εδώ έχω καμιά απόδειξη και νομίζω ότι πολλοί δρούν εδώ και αντιδρούν στην βάση φημών. Είναι σημαντικό λοιπόν να παρακολουθούμε τα γεγονότα, αλλά βεβαίω να βασιζόμαστε σε αντικειμενικά στοιχεία και γεγονότα. Μάλιστα, η κυρία Χόλμαερ. Εκπλήσωμαι κάπως, το ομολογώ, διότι συνήθως και σοσιαλιστές δημοκράτες αλλά και άλλες πολιτικές ομάδες δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο όταν ε, στοχεύουν μια συγκεκριμένη χώρα. Εγώ δεν το πράττω αυτό. Σημειώνω ωστόσο κάτι. Πρώτον, απευθυνόμενοι στον κύριο Μποστινάρου. Δεν ήταν η κυρία Μακοβέη αυτή που ζήτησε τη σύγκληση της ε, συνεδριάσεως. Ήταν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής που απίθυναν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής μας, ο οποίος μετά προσεκάλεσε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, βεβαίως, τίθεται εδώ ένα ερώτημα εφόσον εξετάζουμε την υπόθεση Πόντα, το ερώτημα είναι εδώ η ρουμανική δικαιοσύνη έχει την δυνατότητα να προβεί σε έρευνες για τον κύριο Πόντα ή παρακολύεται στις έρευνες αυτές λόγω του ότι δεν έρεται η ασυλία του κυρίου Πόντα. Αυτά βεβαίως απασχολούν ως γενικό ερώτημα, ανεξαρτήτως πόντα, ανεξαρτήτως το όνομα του πόντα, σε κάθε τέτοια περίπτωση. Θα πρέπει να εξετάζεται η νομοθεσία που αποτελεί την βάση για τα πράγματα αυτά. Δεύτερο, για τα 23 νομοθετήματα, η ταχύτητα με την οποία πρόκειται να ψηφιστούν και να εγκριθούν τα νομοθετήματα αυτά, όντως είναι εκπληκτική διότι τίθεται και ερωτήματα όπως τα συγκεκριμένα μέτρα θα επιτρέπονται μόνο εφόσον είναι απολύτως πέραν πάσης αμφιβολίας άρα δηλαδή διαδικασίες στη βάση απλών ενδείξεων δεν θα είναι πλέον παραδεκτές. Δεύτερο παράδειγμα. Μάρτυρες που αξίζουν της προστασίας δεν θα προστατεύονται στο μέλλον. Γνωρίζουμε τη διαδικασία αυτή και από τις διώξεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Τέτοια νομοθετήματα θέτουν σοβαρά ερωτήματα. Πρέπει να εξεταστούν και πρέπει να κριθούν τα νομοθετήματα αυτά. Το ίδιο ισχύει και για θέματα όπως Εάν στο μέλλον, σε αντίστοιχες διαδικασίες, όπου πρόκειται για υποθέσεις διαφθοράς, μπαίνει μια προθεσμία έξι μηνών, όπου πρέπει να γίνει καταγγελία. Άλλα ερωτήματα. Τα αναφέρω ενδεικτικά. Ερωτήματα, έτσι. Δεν εκφράζω προσωπική κρίση, θέτω ερωτήσεις. Και μεταξύ αυτών των ερωτήσεων συγκαταλέγω και την εξή ότι εκτιμάται οι πορισμένες περιστάσεις να προβλέπονται υποχρεωτικά ποινές κατά δικαστών και εισαγγελέων εάν η διάρκεια της διαδικασίας ή εάν διαπιστώσει παραβιάσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορεί σε μια διαδικασία να προκύψουν και σφάλματα. Αυτό μπορεί να συμβεί παντού. Και τότε στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η δίωξη δικαστών και εισαγγελέων. Επιθυμώ να τεθούν τα ερωτήματα αυτά για λόγους ουσιαστικούς. Ας πάψουμε να συμπαρατασσόμεθα σοσιαλιστές με σοσιαλιστές και χριστιανοδημοκράτες με χριστιανοδημοκράτες, Το πρόκειται δηλαδή για την προστασία των οικείων κυβερνήσεων. Έχουμε ουσιαστικά θέματα, ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ το έπραξα αυτό και στην περίπτωση τη Ουγγαρίας. Ας λάβουμε απόσταση από αυτά τα πράγματα. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνη, δημοκρατία, αρχή του κράτους δικαίου, σεβασμό των κριτηρίων της Κοπενχάγης και στην περίπτωση τη Ρουμανίας, όπως και στην περίπτωση τη Ουγγαρίας. Να κριθούν με τον ίδιο αντικειμενικό τρόπο. Και παρακαλώ και τι και του συναδέλφου τη σοσιαλιστική πλευρά να συμμετάσχουν με εκπλήσει δε το γεγονό ότι ορισμένοι άλλοι δεν ζητούν καν τον λόγο, ενώ μέχρι τώρα ήταν λαλίστα σε άλλε παρόμοιε περιπτώσει. Εγώ τονίζω ότι, λέει, στον ίδιο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Α, θα τα πω στα γερμανικά. Εάν υπάρχουν κατηγορίες, οφείλουν να διερευνηθούν. Να κάνετε τώρα, σαν εμείς να αποτρέπουμε οποιαδήποτε διερεύνηση της αλήθειας, αυτό το βρίσκω ανήκουστο πραγματικά. Α, δεν είπα αυτό όλοι κύριε Χολμαϊρ. Ελπίζω να μπορέσετε τελικά να ψηφίσετε. Όχι, αγαπητή Μπίρκετ Τσίπλη, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μην ισχυρίζετε τέτοια πράγματα. Εγώ είπα ακριβώ το αντίθετο. Παρακάλεσα μάλιστα να αποστασιοποιηθούμε οποιασδήποτε πολιτικέ τοποθετήσει. Να θέσουμε τη συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αφηρημένο, δηλαδή πέραν συγκεκριμένων περιπτώσεων. Είμαι... Η καλοσύνη μου με οδήγησε να δώσω δύο λεπτά έξτρα στις συντονίστριες, ίσως το μετανιώνω τώρα αυτό. Λέει ο πρόεδρος. Πάντω νομίζω ότι διατηρήσαμε μια δικαιοσύνη στην κατανομή του χρόνου. Α παραμείνουμε σε αυτά. Έχουμε λίγο χρόνο για τον ε, πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο ο καημένο περιμένει υπομονητικά για να μπορέσει να σα απαντήσει. Σα παρακαλώ κύριε αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα-δύο λεπτά να σα δώσω ε, το ιστορικό μου με την Ρουμανία. Θυμάμαι πάρα πολύ όταν ήμουν νεαρό διπλωμάτη ακόμα και πήγα στις αρχές των 90, τέλη του 80 στη Ρουμανία. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ακόμα και ζωντανά είναι στη μνήμη μου πώς η χώρα αυτή υπέφερε από ένα σύστημα το οποίο ήταν τόσο φρικτό ώστε κανείς δεν μπορούσε να αναπτύξει το προσωπικό του δυναμικό, να ανθίσει. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πόσο ε, ήταν οι άνθρωποι σε ανέχεια και προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Και επίσης θυμάμαι πάρα πολύ ζωηρά ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ε, μπορούσα, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, να γράψεις τα παιδιά σου στο σχολείο ή ε, αν δεν σε βοηθούσε το κόμμα ή αν δεν λάδωνες έστω και πιο, ε, το πιο χαμηλό ε, δημόσιο υπάλληλο. Το, αυτή είναι η Ρουμανία του τότε και η Ρουμανία του σήμερα είναι μια εκβάθρον διαφορετική χώρα. Και καλό θα ήταν και δίκαιο να μην κάνουμε μία φωτογραφική καταγραφή της κατάστασης σήμερα και να στιγματίζουμε τα κακό κείμενα που μπορεί να είναι πολλά, αλλά να σημειώνουμε και τι έχει επιτευχθεί την τελευταία 25 ετία που είναι αξιοσημείωτα και αξιοθαύμαστα τουλάχιστον. θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας αυτό γιατί έχουμε τόσες μεγάλες ε, δυσκολίες. Ο κύριος Σόγκαρ Αναφέρθηκε στις εθνικές μειονότητες. Υπάρχουν ζητήματα, αλλά προσωπικά ε, είχα και με τον Μαξ Βαντερστούλ ε, στην Τρανσιλβανία εμπειρία που ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση με τις εθνικές μειονότητες. Βεβαίως και παραμένουν τα προβλήματα, αλλά αν συγκρίνεται με την τότε κατάσταση έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Και θα πρέπει να πω και να ευχαριστώ ε, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα θεσμικά όργανα και τη βοήθεια που παρέχουν εκεί. Τα πάντα λοιπόν εντάσσονται σε μία προοπτική και εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει κανεί. Και ένα πολιτικό κόμμα όπως το Ούντεμερέ ε, συμμετείχε ανεξαρτήτως ε, κυβέρνησης σε όλες τις κυβερνήσεις. Και ε, είναι και θετική εξέλιξη αυτή για τις μειονότητες. Ε, τούτων εξέντων βεβαίως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, αν το είχαμε δεν θα υπήρχε αυτός ο μηχανισμός για τη συνεργασία και την επαλήθευση. Ε, και δεν έχει τελειώσει αυτή η προσπάθεια. Θα πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια για να ολοκληρώσει το έργο της και να ε, φτάσουμε ε, σε ένα οριστικό αποτέλεσμα που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση Πόντα έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα πρόοδου. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, όχι. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το είπα πάρα πολύ ξεκάθαρα στον πρόεδρο της Γεωρουσίας. Του είπα ότι πιστεύω ότι σε ένα κράτος δικαίου δεν έχει νόημα να επιτίθεται κανείς ε, προσωπικά στον πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και το έκανε ο ίδιος και του τόπο προσωπικά, ότι αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα ε, προς επίλυση to, to maintain. και ε, θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για το κοινοβούλιο, για την ασυλία. Κάθε κοινοβούλιο έχει κάποιο σύστημα ασυλίας για τα μέλη του. Αλλά θα πρέπει να πω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, η ασυλία σχεδόν σε όλα τα κοινοβουλευτικά συστήματα στον κόσμο συνδέεται με τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες του κάθε προσώπου για να προστατεύουν τον βουλευτή στο βουλευτικό του έργο και δεν θα πρέπει να επεκτείνονται επέκεινα αυτού. Και το έχω πει και στους δύο πρόεδρους και των δύο σωμάτων της Βουλής ότι εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την ασυλία και θα κρυθούν οι πάντες και υπό το φως αυτό και υπό το πρίσμα αυτής της αρχής. Δεύτερον, αν ληφθεί η απόφαση της ασυλίας και όταν λαμβάνεται αυτή θα πρέπει να βασίζεται στα ίδια κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ε, δικάζονται και οι υπόλοιποι πολίτες ενώπιον των δικαστήριων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση ε, αν είσαι εκλεγμένος βουλευτής ή όχι. Αυτή τη στιγμή σε έχει αρθεί η ασυλία σου. Αυτά ισχύουν και για τις τροποποίησεις των νόμων όταν εγκριθούν αυτά τα νομοσχέδια. Και συμφωνώ με την κυρία Σίπελ, ποιος το είπε δεν ξέρω, ο κύριος Νίντερ όταν λέγει ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στη συζήτηση στο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Αυτό μας έλειπε. Είπαμε, ε, θα πρέπει να σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά και της νομοθετικής εξουσίας. Αλλήμον. Το λέμε όμως και αυτό. Σε περίπτωση που εγκριθεί το α ή το β, ενδεχομένως μπορούμε να καταλήξουμε στο α ή β συμπέρασμα απάντησα σε μια γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση για ε, κάποια νομοσχέδια στη Γαλλία και τους είπα αν περάσει αυτός ο νόμος θα μπορούσε να θέσει τα εξή ζητήματα. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και στην παρούσα περίπτωση. Ξέρετε, καμιά φορά και πρακτικά και πολιτικά είναι πιο ευφυές να προειδοποιείς ότι πρόσχε αυτό το δρόμο που έχεις πάρει μπορεί να είναι στραβός. Αντί να περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν νόμος και να χρειαστεί στη συνέχεια τροποποίηση αυτού του νόμου και αναθεώρηση της νομοθεσίας. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια τέτοια ισορροπία. Για την ακαιρεότητα των πολιτικών ηγετών. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να τεθεί πολύ γενικά αυτό το ερώτημα, αλλά όταν τίθεται, γίνεται συγκεκριμένο, δεν είναι γενικό, γιατί όλοι ξέρουμε περί τίνος πρόκειται για τον Πρωθυπουργό ε, Πόντα ε, και ε, την δίωξή του. Η κυρία Σίπελ σωστά είπε ότι η έρευνα αφορά κάποιες κατηγορίες και αιτιάσεις στο διάστημα πριν εκλεγεί. Έτσι, αυτό είναι γεγονός, είναι αντικειμενικό γεγονός και επιβεβαιώνεται. Είναι όμως σαφές. Μπορεί να λες από τη μια ότι οι βουλευτές και οι πολίτες, οι πολιτικοί και τα δημόσια πρόσωπα δεν θα πρέπει να έχουν πιο ευνοϊκή μεταρρύθμιση από ότι οι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και εμείς να ε, δίνουμε το παράδειγμα, να έχουμε υψηλότερες προδιαγραφές και πρότυπα. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής ηθικής. Δεν είναι νομικό ζήτημα και το συμμερίζεστε πιστεύω ευρέως και στο Κοινοβούλιο αυτό. Αυτό τον έφερα. Δεν είναι εθνικό ζήτημα και συμφωνώ, είναι ευρύτερο, αλλά θέλω να το θέσω και στο πλαίσιο αυτό του μετασχηματισμού που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω. Έχουν επιτευχθεί ήδη πάρα πολλά, αξιοσημείωτη, αξιοθαύμαστη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή ώστε να μην είναι αναστρέψιμη, αλλά όταν συγκρούονται δύο εξουσίες, ιδιαίτερα η νομοθετική και η δικαστική και ανοιχτά ε, επικρίνονται και αλληλοκατηγορούνται, δεν είναι καλό, δεν είναι, είναι προς τιμή κανενός. Ε, και ελπίζω αυτό οι πάντες να το κατανοούν και στη Ρουμανία. Ταυτόχρονα όμως είναι γεγονός ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί ελεύθερα σε όλα τα επίπεδα και να μην αυτοπεριορίζεται. Μου ζήτησε η κυρία Γκόμες να είμαι σκληρός. Εγώ δεν έχω τη φήμη ότι είμαι ιδιαίτερα επίκης. Ε, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε αυτό σας το αίτημα. Και σήμερα, α, κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω στην κυρία Χολμάιερ ότι όταν επικρίνουμε ηγέτες, πολιτικούς, πρωθυπουργούς, δεν επικρίνουμε τις χώρες, πρόσωπα και πολιτικούς επικρίνουμε. Οι χώρες δεν είναι πολιτική τους και το λέω ως πολιτικός και πάλι καλά δηλαδή. Για το ε, θέμα των σκύλων, ε, των αδέσποτων, ξέρω ότι αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Ε, Πολλοί κόσμος ανησυχεί στην Ευρώπη και φαίνεται ότι είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με τα αδέσποτα σκυλιά στη Ρουμανία. Αλλά επειδή εγώ λατρεύω τους σκύλους και έχω και σκύλο, πρέπει να σας πω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν έχεις ένα παιδί στο δρόμο που πεθαίνει επειδή το δάγκωσε ένα δέσποτο σκυλί, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος αν δεν κάνεις τίποτα για να τα μαζέψει ο Μπόγιας. Το ξέρω ότι θα πρέπει να είναι ανθρώπινη μεταχείριση και ε, σωστή και φυσικά χωράει πολύ βελτίωση εκεί, αλλά ε, είναι δύο οι πλευρές της ιστορίας αυτής, δεν είναι μία. Και θα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο γιατί έχουν συμβεί και ανθρώπινα δράματα και σοβαρότατα λόγω των αδέσποτων σκύλων, όχι μόνο στη Ρουμανία, αλλά και στη Ρουμανία. Και τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε, γιατί ξεπέρασα και το χρόνο μου, είναι το εξή. Εγώ χάρηκα που έγινε αυτή η συζήτηση, πραγματικά, ειλικρινά, ήμουν πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας και φανταζόμουν ότι θα ήταν ε, πολιτικά ορμόμενη αυτή η προσπάθεια το ένα κόμμα κατά του άλλου, αλλά ε, με εξεπλάγει ε, ευχάριστα και θετικά από το γεγονός ότι η Επιτροπή σας ήθελε να συζητήσει τα δομικά ζητήματα και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να λυθούν αυτά. Και θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και θα το πω ότι διακομματικά συμφώνησε η Επιτροπή σας ότι η Ρουμανία έχει επιτελέσει μεγάλη πρόοδο σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την υπομονή σας. Um, σας ευχαριστώ ε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής βλέπετε σας χειροκροτούν και όλα οι συναδελφοί μου και ευχαριστώ και εσάς ε, συναδελφοί. Ξέρω ότι θέλετε να φύγετε. Μιλήσατε για ε, ένα είδος συνωμοσία δίθεν της μιας ε, πολιτικής ομάδας κατά της άλλης αλλά και χαρήκατε που δεν συνέβη ε, αυτό στην πραγματικότητα είναι ένας μηχανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουμε μέσα εδώ στην Επιτροπή μας πολύ σκληρός μηχανισμός έχουμε ένα μηχανισμό εμείς είναι δυναμική ιστορία δεν είναι στατική και βέβαια προκαλεί εντάσεις όπως ε, προκάλεσε σήμερα. Τα συζητούμε αυτά βέβαια διαρκώς. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τις και τους συναδέλφους που καταφέραμε και ξεπεράσαμε ε, τον κάβο αυτόν με πειθαρχία και ηρεμία. Είναι δύσκολο θέμα, αλλά είναι και ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον εξετάζουμε τι συμβαίνει στην κάθε χώρα μέλος. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής μου και ευχαριστώ και εσά κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπή που προσήρθατε και μας απαντήσατε με καλή διάθεση και με αρκετή ακρίβεια. Ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε ξανά τα θέματα αυτά εφόσον το επιθυμείτε στη συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σα και αποχαιρετώ τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Colleagues, we uh, move straight to the next. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το υπαριθμόν 8, γιατί έχουμε, βρισκόμαστε σε κάποια καθυστέρηση. Μήπως μπορείτε ε, να μετακινηθείτε εκτός εθούσης εάν δεν πρόκειται, αν δεν επιθυμείτε να παραμείνετε. Η συγητή συγγνωμοδοτήσεως είναι ο κύριος Νίντερ Μούλερ και προβλέπεται και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φερνάντες, τον εισηγητή δηλαδή του προϋπολογισμού του 2016. Να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Νίτερ Μούλερ για τις ε, προτεραιότητες μας για το 2016. Το θέμα είναι σημαντικό. Αν δεν σας απασχολεί τόσο πολύ, παρακαλώ εξέλθετε τις ερωτήσεις και θα παρακαλέσω τον κύριο Φερνάντες ε, να σχολιάσει τις προτεραιότητες της Επιτροπής ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών. Κύριε Φερνάντες, εσείς λοιπόν πρώτος. Α, όχι, διακόπτει ο κύριος Μωράς. Ο κύριος Νίντα Μιλά. Με συγχωρείτε κύριε Φερνάντες, ο κύριος Νίντα Μιλά. Πέτερ εσείς. Στα αγγλικά. Δεν ακούω τη φωνή μου, αλλά ναι. Έκανε λάθος, ε, παραδέχτηκε ο πρόεδρο κ. Μωράε και έδωσε το λόγο στον κ. Φερνάντε πρώτα. Σας παρακαλώ πρώτα εσείς κύριε, Νίτερ Νίντερ Ευχαριστώ τον ε, κύριο Φερνάντες που είναι σήμερα παρόν και θέλω να αναφερθώ σε ορισμένες προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τον προϋπολογισμό του 2016. Από τις προτεραιότητες αυτές, ορισμένες έχουν περιληφθεί σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος μας Μωράες στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γενικά το πρώτο θέμα ανάγεται στην τρέχουσα συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές μέσω της Μεσογείου και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ροές αυτές. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό για μας. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προτεραιότητες που θέλω να υπενθυμίσω εδώ. Πρώτα, αύξηση στα ταμεία ασύλου, μεταναστεύσεως κλπ. για να διασφαλιστεί ότι η επανεγκατάσταση, ο μηχανισμός δηλαδή επανεγκατάστασης και μετακίνησης να είναι πραγματικά χρηματοδοτημένοι για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ε, προσφύγων, μεταναστών, ε, ετούντων άσυλο κλπ. Δεύτερο, επαρκής χρηματοδοτική ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μεσόγειο, ιδίως για ε, επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης. Επίσης να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ασων για το προσωπικό και για τη λειτουργία του για το 2016 για λόγους τεχνικούς. Μας ικανοποιεί η προτινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού Frontex για τις επιχειρήσεις τρίτων και ποσειδών, αλλά ιδίω για να διασώζονται οι ζωές των ανθρώπων στη θάλασσα. Πρέπει να είναι ο βασικός στόχος αυτών των επιχειρήσεων. Για τους οργανισμούς η Επιτροπή ε, Θεμελιδών Ελευθεριών επαναλαμβάνει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επανεξετάσει τα σχέδιά της για να λάβει καλύτερα υπόψη τον φόρτο εργασίας των διαφόρων οργανισμών. Για το τελευταίο θέμα ζητούμε βελτίωση του, της χρηματοδότησης για δράσεις προώθησης του κράτους δικαίου. Εκτός από αυτές τις βασικές προτεραιότητες θέλω να σας ε, ρωτήσω και για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Φερνάντες, για την απόφαση για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Όπως θα γνωρίζετε, η χρήση του μέσου ευελιξίας συναποτελεί μέρος της προτάσεως της Κομισιόν για έναν επίγοντα μηχανισμό μετεγκαταστάσεως για να ενισχυθούν η Ελλάδα και η Ιταλία η Επιτροπή Προπολογισμών πώς θα αντιμετωπίσει την πρόταση αυτή εκ παραλίλου με, το, με διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού 2016 επειδή η προτινόμενη αύξηση αναφέρεται στον προϋπολογισμό 2016 ή θα προωθηθεί ταχύτερα μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τον Relocation Mechanism. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά είναι πολύ χρήσιμα αυτά που είπατε και βεβαίως θέσατε ξεκάθαρες ερωτήσεις στον αγαπητό Φερνάντε, τον οποίο θα παρακαλέσω τώρα να σχολιάσει τις προτεραιότητες αυτές της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Κύριε Φερνάντες, επιθυμείτε να σχολιάσετε τις προτάσεις ε, Νίντερ Μιούλερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι να σας παρουσιάσω τις ε, γραμμές προσανατολισμού που έχουν ήδη ψηφιστεί. Έχουν ψηφιστεί και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού η έκθεση για την εντολή και για τον τρίλογο για τις γενικές μας προτεραιότητες. Να θυμίσω ότι στις 11 Μαρτίου ψηφίσαμε για τις κατευθυντήριες γραμμές και σε αυτές ε, στηρίξαμε τα τρία ε, απασχόληση, δηλαδή αμπλουά, επιχειρηματικότητα, ε, και αλληλεγγύη και αλληλεγγύη στη, στη μετανάστευση. Και βεβαίως αυτές οι προτεραιότητες έχουν στη συνέχεια δημοσιονομικές επιπτώσεις στις αντίστοιχες γραμμές για τα προγράμματα. Ξεκινάμε από μια αρχή. Την αρχή στον προϋπολογισμό μάλλον του 2016, ότι δηλαδή οι δεσμεύσεις μας ε, θα πρέπει να ε, τηρηθούν. Δηλαδή οι ε, δέσμευση του Συμβουλίου απέναντι στο Κοινοβούλιο και αρχίζω την απάντησή μου για την ευελιξία. Δέσμευση του Συμβουλίου σε σχέση με το πολιετές σε δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να πούμε ότι είναι διαφορετικό Όσο ό,τι αφορά την ευελιξία από το πλαίσιο του 2007-2013, το δεχτήκαμε μειωμένο γιατί έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία. Τι είναι η ευελιξία? είναι διάφορα μέσα ευελιξίας και έχουμε συμφωνίες με το Συμβούλιο γιατί τα μέσα ευελιξίας όπως ας πούμε το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα μέσο ε, ευελιξίας και πρόκειται για μέσα τα οποία βρίσκονται άνω του δημοσιονομικού πλαισίου του PDP Και έχουμε επίσης και τα αποθέματα, που, τα αποθεματικά που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο χρόνο, από το 2016 θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για τις υποχρεώσεις. Γιατί πάνε σε ένα γενικό αποθεματικό. Με έναν μικρότερο προϋπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και για λόγους αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φιλονευελιξία και αυτά τα μέσα ευελιξία. Να σεβαστούμε τις δεσμεύσει. Και αυτό είναι κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το πρόβλημα των πληρωμών. Είναι απαράδεκτο να έχουμε πάνω από δύο δις ε, καθυστερήσεις. Είναι ανεξόφλητος λογαριασμός. Είναι ε, τρελό. Και θα πρέπει το Συμβούλιο να πληρώσει τα χρέη του τα ζωγαριασμό του. Αυτά τα οποία ανέκρινε, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Είναι απαράδεκτό να γίνεται αυτό και μάλιστα σε σημαντικές κατηγορίες. Κατηγορία 3 δεν έχει αποθηματικό. Αυτό θυμίζει ότι έχουμε πρόβλημα. Για παράδειγμα, για τα πιλωτικά σχέδια ή για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι 124 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση για το μέσο ευελιξίας, αλλά δεν αρκεί κατά τη γνώμη μας, γιατί Γιατί θέλουμε μεν αυτό το, το αποθηματικό, αλλά θέλουμε και για τις πιλωτικές δράσεις και για τις παρασκευαστικές δράσεις. Τώρα, Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό για τούτην εδώ την Επιτροπή, έχουμε αυξήσει για δύο ταμεία, τα κύρια ταμεία, το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση, την ένταξη, το ΜΙΦ, ε, αύξηση των υποχρεώσεων κατά 36,3% που είναι σημαντικό και έχουμε 7,5% αύξηση των υποχρεώσεων ε, στο Ταμείο το Ταμείο Ασφάλειας. Και αντίστοιχα έχουμε το ίδιο και για τις πληρωμές. Για τα προγράμματα δικαιοσύνη και το πρόγραμμα, το πρόγραμμα ισότητα δικαιωμάτων του πολίτη έχουμε αύξηση και ταυτόχρονα συγκρίνω με το 2015 έχουμε μια αύξηση της τάξης του 4,5% στις υποχρεώσεις. Έχουμε ακόμα κάτι γενικό για τον τριμερή διάλογο. Το 5% μείωση του προσωπικού τα επόμενα πέντε χρόνια άρα δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί το ίδιο και για τους οργανισμούς που δεν είναι όλοι οι ε, ίδιοι. Έχουμε κάτι επίγον. Όταν μιλάμε για τους οργανισμούς, βλέπουμε πούμε ότι το Frontex ε, έχουμε αύξηση στις ε, υποχρεώσεις 3-4% ενώ έχουμε το σοργαν... την Ιάζο για μείον 4% ενώ το ευρωπαικο οργανισμο για τη Δικαιοσύνη και τα Θεμολιώδη Δικαιώματα ε, μείον 4%. Πρόκειται για οργανισμού που δεχτήκαμε γιατί είναι οι προτεραιότητέ μα Έχουμε βάλει στην έκθεσή μα για την εντολή μια γενικότερη ε, μέρημνα για τους οργανισμούς αλλά και πιο συγκεκριμένη μέρημνα όσον αφορά τον οργανισμό, τον οργανισμό στήριξης για το άσυλο και την Europol που τελικά αφορούν την ε, ΛΥΜΠΕ. Πρόσφατα υιοθετήσαμε το διορθωτικό σχέδιο προπολογισμού αριθμός 5 θα ψηφιστεί στην επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου. Η Κομισιόν προτείνει ενίσχυση 16 θέσεις για το Frontex, 4 για την EASO και 3 θέσεις για την Europol. Αλλά μετά είναι κάπως γελίο γιατί λόγω του κανόνα του 5% στην πρόταση σχεδίου προπολογισμού για το 2016 της Κομισιόν έχουμε λιγότερες θέσεις για το Frontex, λιγότερες θέσεις για την Europol και μείον τέσσερι θέσει για την Eurojust. Πράγμα που αποδεικνύει αυτό που έλεγα, ότι πρέπει να αναλύσουμε αναπερίπτωση τα θέματα προσωπικού για τους οργανισμούς. Να θυμίσω κάτι ακόμα. Ότι μιλάμε για ένα σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν, για ένα σχέδιο προπολογισμού που το Συμβούλιο θα κάνει μια ανάγνωση και, και κανονικά περιμένω ακόμα τα, χειρότερο, τα χειρότερα από την ανάγνωση εκεί. Γιατί το Συμβούλιο κάνει ωραίες δηλώσεις και τις δεχόμαστε και συμφωνούμε, αλλά μετά, στη συνέχεια, το χρήμα δεν ακολουθεί κάποιες φορές ούτε καν τα χρήματα για να πληρωθούν ε, τα όσα έχουν ήδη τελειώσει δεν δίνει, όπως σας είπα. Οπότε θα διαπραγματευτούμε με αυτές τις προτεραιότητες που ανέφερα. Έχουμε προτάσεις και σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν με αυξήσει, αλλά και επικρίσεις που είναι σαφείς στην παρέμβαση που ήδη κάναμε. Τώρα θα έχουμε επίσης ε, εντολή για τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Μετά το Σεπτέμβριο έχουμε την προθεσμία κατάθεσης για τις δημοσιονομικές ε, μετα... Ε, τροπολογίες και αυτό θα είναι πιο συγκεκριμένο γιατί σε αυτή την έκθεση για την εντολή δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα διευκρινίζουμε μόνο τους οργανισμούς ε, ε, που σας ανέφερα. «28-30 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε για αυτές τις τροπολογίες. Το με Σεπτεμβρίου για την ε, το κείμενο και τον Νοέμβριο έχουμε τη σύνοδο που θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό. Εγώ αναμένω το Συμβούλιο να τηρήσει τις υποσχέσεις του και ότι οι πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες έχει ανακοινώσει να μεταφραστούν σε δημοσιονομικές υποχρεώσεις και πληρωμές. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Και τώρα θα πάρουν το λόγο οι Σκιώδης. Ο Τόμας. Ε, μετά ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με ευχαριστίες. Για το, ε, προς το Πέτερ για τον τρόπο με τον οποίο έκανε ε, τις διαπραγματεύσεις και τις συνεδριάσεις με τους και ηγητές που ήταν πάρα πολύ επικοδομητικές. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ένα έχω να πω. Θέλουμε να δούμε αύξηση για ε, το Frontex και τον άλλο οργανισμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις. Frontex, EASO, Europol και Eurojust θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον κανόνα ε, της μείωσης του προσωπικού, που είναι μια υποχρέωση που αφορά όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την πολιτική μας αυτή της μείωσης του προσωπικού, διότι έχουμε αυξημένα καθήκοντα πλέον ε, στους συγκεκριμένους οργανισμούς. Δεν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα και το έχουμε συζητήσει. Περισσότερα καθήκοντα με λιγότερο προσωπικό. Επίση θέλουμε αύξηση στον προπολογισμό ΕΑΣΟ και Ευρωπόλ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές από τη μετανάστευση και να καταπολεμήσουν ε, αποτελεσματικά την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι για πολύ καιρό τώρα δεν έχουμε αυξήσει τα κονδύλια στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Και θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας τα τελευταία έξι χρόνια έχουν σχεδιαστεί πάνω από 15 νέα συνθετικά ναρκωτικά. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, λοιπόν, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξανασκεφτεί αυτό και πάρα πολύ προσεκτικά. για τις ανάγκες του MCDDA που είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή, πιστεύω. Θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο στρούθο καμιλισμός για τα ναρκωτικά. Και έχει οξυνθεί η κρίση αυτή με τα ναρκωτικά λόγω και της οικονομικής κρίσης. Σταματώ εδώ, όλα τα υπόλοιπα υπόθηκαν ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους για την επικοδομητική του στάση. Ευχαριστώ Τόμας. Ο Κάρλος Κόγιο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω απλά να πω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φερνάντο που έκανε σπουδαία δουλειά όπως έκανα και για το θέμα του σχεδίου Juncker και έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ελπίζω ότι θα σημειώσετε το εξή, κύριε Φερνάνδες, ότι έχουμε έναν προπολογισμό που δεν αρκεί για να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περισσότερη Ευρώπη ενώ να έχουμε έναν ε, κακομήρικο προπολογισμό. Πρώτον. Δεύτερον, στη δική μας Επιτροπή έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, όπως μάλιστα σωστά αναφέρθηκαν από τους δύο ομιλητές που προηγήθηκαν και από τον αγαπητό Τόμας. Έχουμε μπροστά μας το θέμα της Μεσογείου, την πίεση των μετανάστευσης, το σετώντες ε, άσυλο και έχουμε ένα τεράστιο κύμα όπου δεν έχουμε μέσα και απαντήσεις. Και αν κάποιες απαντήσεις μπορούμε να τις προβλέψουμε στον προπολογισμό και δεν είναι και προφανές ότι λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την εκδοχή που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, πάντως σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα όπως ε, το μηχανισμό ευελιξίας όπως είπε ο συνάδελφος Νίτερ Μούλερ. Και, και σωστά τα είπε. Πρέπει να ε, μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πήγουσες ανάγκες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι λόγω διαδικασίας δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Και τρίτον, και ο κύριος Φερνάντο τον, ανέφερε έφερε αυτό, ότι συχνά η σχέση στην εκπόνηση του προπολογισμού οδηγεί ότι το Κοινοβούλιο μόλις μπορεί να αποκαταστήσει τις προτάσεις της Κομισιόν. Δηλαδή η Κομισιόν κάνει την πρόταση, το Συμβούλιο μειώνει το κονδύλια και το κοινοβούλιο ξαναβάζει τα αρχικά κονδύλια. Όμως ούτε αυτό δεν αρκεί κάποιες φορές. Οι φετινές προτάσεις ήταν κάτω από τις πραγματικές ανάγκες. Ο Τόμας ε, σωστά και μόλις τελείωσε να λέει ότι ε, ε, το παράδειγμα του οργανισμού καταπολέμησης του ναρκωτικών. Η ιδέα ότι πρέπει σε όλους τους οργανισμούς να εφαρμόσουμε ένα, μία μείωση προσωπικού της 65% μπορεί να έχει νόημα στους μεγάλους οργανισμούς, αλλά στους μικρούς ε, μία μόνο θέση, κατάρριξη μόνο μία θέση, μπορεί να σημαίνει ότι μία ουσιαστική λειτουργία θα πάψει. Γιατί σε αυτούς τους μικρούς οργανισμούς το να βγάλεις ένα κομματάκι δεν πρόκειται να βοηθήσει στον προπολογισμό της Ένωσης, αλλά μπορεί να βλάψει, να ζημιώσει σημαντικά τη λειτουργία του εν λόγω οργανισμού. Ελπίζω πως θα μπορέσετε κύριε Φερνάντες να διαβιβάσετε αυτή την ευαισθησία της Επιτροπής μας στην Επιτροπή Προπολογισμού. Πρόεδρος, δεν θέλω να περικόψω τη συζήτηση για τον προπολογισμό, γιατί είναι μια από τις πιο σημαντικές που κάνουμε εδώ, αλλά ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κλείσουμε ε, γρήγορα, γιατί έχουμε και την ακρόαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους υποψηφίου. Και πρέπει να την κάνουμε απόψε. Γι' αυτό και ζητώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Και εσείς συνάδελφοι, συγγνώμη που σας πιέζω. Ε, έχεις το λόγο. Ναι, θα τα πω όμως σου ειδικά. Ίσως τα σου ειδικά να τα πω πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε απολύτως όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό που να βοηθάει στη διάσωση των ζωών και των ανθρώπων. Δεν θέλουμε την καταστολή, θέλουμε οι πόροι να πηγαίνουν στα κράτη-μέλη που χειρίζονται υπεύθυνα. Εσείς ζητάτε περισσότερα χρήματα ε, για τον ΕΑΣΟ, αλλά εμείς επαναλαμβάνω δεν πιστεύουμε στα κατασταλτικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ολιστικό έδαφος. Τα κράτη-μέλη τώρα ε, απορρίπτουν την πρόταση για ε, επανεγκατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών και προτιμούν κατασταλτικά μέτρα. Λεφτά για στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκουμε για να πυροβολούμε τα σκάφη με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εμείς θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αλλού για την επανεγκατάσταση ε, των προσφύγων. Στο προπολογισμό του 2016 θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση και αν δεν μπορεί να το κάνει το Συμβούλιο θα το κάνουμε μόνοι μας. Πάντα είστε σύντομοι, είτε μιλάτε σουηδικά είτε μιλάτε αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το συγγνώμη που σε πιέζω. Πείτε πρώτα και μετά ο κ. Φερνάντες. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι πραγματικά εξαιρετικά σύντομο. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντε. Σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα και τι παρατηρήσει σα. Ευχαριστώ και τους και Συμφωνώ Συμφωνώ, Τόμας. Είχαμε πολύ καλή ατμόσφαιρα ε, στην ομίγυρη των ε, σκιωδών. Θα συνεχίσουμε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τον προπολογισμό του 2016. Ευχαριστώ. The ο κύριος Φερνάντες. Όντως ο προπολογισμό μας είναι μικρός, είναι σχεδόν το 1% του ε, ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ε, της Ένωσης. Ένας προϋπολογισμός που δεν επιτρέπει ε, να εξυπηρετήσουμε όλες τις προτεραιότητες και όλες τις νέες αρμοδιότητες. Είναι βεβαίως 145 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι σημαντικό για την Ευρώπη το ποσό αυτό και έχει μεγάλη προσθέμενη αξία. Θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους Ευρωπαίους ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι 94% για επενδύσεις και μόνο 6% διοικητική λειτουργία που σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικός προϋπολογισμός, έχει μια μεγάλη όπως είπα προσθέμενη αξία που όμως χρειάζεται νέους ιδίους πόρους. Βεβαίως αυτή είναι μια συζήτηση που δεν θα γίνει εδώ και η διάκριση ανάμεσα σε δικαιούχους και απορρίπτες δηλαδή των κονδυλίων και καθαρές συνεισφορείς είναι μια ερώτηση, είναι μια συζήτηση κακή και οδηγεί στη δίκαιη επιστροφή και σε χώρες οι οποίες είναι σύμφωνες με το δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτικό εκεί, υπάρχει ομοφωνία δηλαδή, μετά όμως προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο, κάνοντας τον και μικρότερο τον προϋπολογισμό εκάστου έτους και από αυτό προβλέπεται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα ίδια κράτη-μέλη που υπερψήφισαν το, δημόσιο, το, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μετά συστηματικά καταψηφίζουν τους προϋπολογισμούς ανά έτος. Δεν λέω ποιες είναι αυτές οι χώρες, αλλά είναι πολλές, δεν είναι μόνο μια. χαμιά. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο που δεν γίνεται ποτέ. Γνωρίζουμε πόσο κοστίζει μια παραπάνω, παραπάνω η απασχόλησης. Θα έπρεπε να γνωρίζουμε πόσο κοστίζει να χαθεί μια θέση απασχόλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι κόβουμε όταν κάτι δεν πρόκειται να κάνουμε. Θα έπρεπε να μάθουμε ποιο είναι το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κοστίζει περισσότερο το, το να μην το κάνουμε θα επαλλάξουμε το όραμα που έχουμε. Να εξετάσουμε δηλαδή το κόστος της παράληψης, της αδράνειας. Βεβαίως, τα χρήματα δεν επαρκούν για πολλούς οργανισμούς, αλλά έχουμε κάποιους περιορισμούς. Ναι, παρακαλώ συντομεύετε. Ναι, έχουμε το δημοσιονομικό πολίτε πλαίσιο. Και επ' αυτού ζητώ την κατανόησή σας. Αν παίρναμε όλες τις τροπολογίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα χρειαζόμασταν ολόκληρο το δημοσιονομικό πλαίσιο για μια χρονιά. Και πάλι δεν θα αρκούσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Μωράες, σας ευχαριστώ πολύ καθώς και τους και οδησίγητες και τον κύριο Νίντερ Μιούλερ. ...15 Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Και τώρα προχωρούμε στο υπαριθμό 11 την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του Προέδρου του FRA, του ε, Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ τα μέλη που προσήλθαν για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Βεβαίως σημειώνω ότι είναι ε, περασμένη κάπως η ώρα, είναι και ε, πέμπτη απόγευμα. Ευχαριστώ πάντως που διαθέτετε τον χρόνο αυτόν για το πολύ σημαντικό άλλωστε θέμα. Έχω κάποιο σημείο μας σχετικά. Sorry, colleagues, I have to some, draw some lots, so I'm just checking. Um... Να εξετάσω μια στιγμή τη διαδικασία, πρόεδρε. Ε, συγγνώμη, συνάδελφοι, με συγχωρείτε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Αν τώρα συμφωνείτε, να προχωρήσουμε τώρα στην ακρόαση για τον διορισμό του, του, του Διευθυντού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού 168 2007 καλούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν την άποψή του και την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων. Υπάρχουν τρει υποψηφιότητε σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού 168-2007 το οποίο άρθρο θεσπίζει ότι στην βάση καταλόγου που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια διαφανή διαδικασία επιλογής καλούνται οι υποψήφοι να απευθυνθούν στο Συμβούλιο και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και μετά τα όργανα αυτά δηλώνουν τις προτιμήσεις τους. Έχουμε υποβάλει ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο στους υποψηφίους με τρεις κοινέ ερωτήσεις. Οι τρεις οι υποψήφοι έχουν απαντήσει γραπτός στο ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις τις βρίσκουν τα μέλη μας στα meeting documents. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Εβδόμου. Θα ψηφίσουμε δηλαδή για να θεσπίσουμε την, ε, την σειρά προτιμήσεων των υποψηφίων. Και τώρα θα κάνουμε κλήρωση για το ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος που θα ακούσαμε. Βεβαίως επειδή είμαστε διαφανείς βλέπετε τα έχω δώσει ένα διαφανές κυπελάκι τα χαρτάκια με τα ονόματα. Ε, είναι διαφανές το κύπελο όπως βλέπετε. Μην τολμήσει κανείς να με κατηγορήσει για προκατάληψη. Δεν γνωρίζω άλλωστε κανένα των υποψηφίων, δεν είναι και συγγενείς μου, ούτε ο παδί μου. Πρώτος ο κύριος Φλάχερτη. Δεν είμαι ούτε Ιρλανδός, ε, κάτι σκοτσέζικο έχω στην καταγωγή μου. Κύριε Φλάχερτη λοιπόν είστε πρώτος. Μετά καταφορετική σειρά, γιατί βέβαια θα μπορούσα να πάρω ένα δεύτερο όνομα. Αλφαβητικά λοιπόν. η κυρία Φαντελάν και η Αμπράνη Κύρις με αυτή τη σειρά. Καλωσορίζω τον κύριο Βράχερτη στην ε, συνάντηση της Επιτροπής Θεμελιωδών Αριστεριών. Ε, να σας πω πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία. Καθίστε κύριε Βράχερτη. Ο υποψήφιος λαμβάνει το λόγο για πέντε λεπτά για ένα κτίριο δήλωση Καλώς ήρθατε στη Λίμπε. Αφού φτάσατε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε και παραπέρα. Μετά από την εισαγωγή σας θα έχουμε χρόνο για την υποβολή 11 ερωτήσεων. Ανά 3 λεπτά. 3 λεπτά δηλαδή για την ερώτηση και 3 λεπτά για την απάντηση. Για τις ερωτήσεις. Θα αναγκαστώ να είμαι πάρα πολύ αυστηρό στην τήρηση των χρονικών ορίων. Οι οι ε, τελευταίοι έσχατοι δηλαδή δεν θα έχουν ε, χρόνο. Σας ε, ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θα τηρήσω το χρόνο για όλους. Έχετε και, έχετε και διερμηνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίσημη γλώσσα εργασίας ε, που επιθυμείτε. Μην μιλείτε πάρα πολύ γρήγορα για να προλαβαίνουμε να σας μεταφράζουμε. Και σα ε, σας υπενθυμίζω ότι θα προβείτε σε μια προφορική τοποθέτηση της τάξης των 5 λεπτών. Είστε έτοιμος? Είστε και εσείς έτοιμες κυρίες και κύριοι? Ε, μην μιλείτε άλλο, δώστε την ευκαιρία στον άνθρωπο να μπορέσει να αναπτύξει τις απόψεις του. Άντε κύριε Βράχαρτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι πολύ μεγάλη χαρά ευκαιρία που έχω να απευθυνθώ σε εσά σήμερα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την έκθεση της ε, Εφράτου Οργανισμού Θεμελιδών ε, Ελευθεριών και Δικαιωμάτων. Ε, είναι βραχή ο βίος του οργανισμού αυτού, αλλά είναι πολύτιμη η δουλειά τους για την προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Όσο προχωρεί λοιπόν αυτός ο οργανισμός θα πρότεινα να βασιστούμε στα επιτεύγματα και στις κατακτήσεις και να επικεντρωθούμε σε τρία σημεία των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Πρώτον, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να ενταχθούν εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, είναι κάθετη η οργάνωση, είναι λίγο σαν σιλό ε, λειτουργούν σε κάποιο πλαίσιο αλλά όχι σε άλλα. Ε, τουλάχιστον σε θέματα ασφαλείας δεν εντάσσονται με το σωστό τρόπο. Το πρώτο λοιπόν είναι το λεγόμενο mainstreaming. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τα κράτη-μέλη να δημιουργηθεί ε, μία συνείδηση, ιδιαίτερα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι κατά κύριο λόγο έργο του οργανισμού. Καλούνται εθνικοί φορείς, τα κράτη-μέλη, να επιληφθούν. Αλλά ε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει πολύ σημαντικό ρόλο ως κέντρο αριστείας για να ε, είναι ως καταλήτης να δράσει τα κράτη-μέλη. Και ο τρίτος τομέας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για μένα έχει να κάνει με εκείνους τους φορείς πέραν των κρατών και του των θεσμών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εδώ σκέφτομαι ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο ο οργανισμός για να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι είναι και δική τους ευθύνη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ας πούμε, η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, η εννέα ψηφιακή αγορά και όλα αυτά τι σημαίνουν και θα κριθεί επιτυχία ε, από μη κρατικού φορείς. Ο Οργανισμός Μελιδών Δικαιωμάτων έχει ως στόχο να σας υποστηρίξει καλύτερα και εδώ και αλλού. Αν με ρωτήσετε γιατί ε, θέτω υποψηφιότητα ή αν έχω τα απαραίτητα προσόντα, να σας πω ποιες ιδιότητες και ποια προσόντα πρέπει να έχει ο διευθυντής. Θα πρέπει να είναι ε, ακρεφνής Ευρωπαίος πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανος πολίτης της Ευρώπης, της Ευρώπης των αξιών, της Ευρώπης που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει εμπειρία ο διευθυντής σε ένα τα πιο δύσκολα έργα. Παίρνεις ένα στεγνό κανόνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κάνεις χειροπιαστή καθημερινή πολιτική νομοθεσία και δράση. Έχω οκταετή εμπειρία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπου ξεκίνησα εντατικό διάλογο με κράτη ανά τον κόσμο ε, για να επιμείνω για τις ευθύνες τους και πραγματικά είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Άλλη ιδιότητα και προσόν που πρέπει να έχει ο διευθυντής είναι η δυνατότητα να κατανοεί την υποστηρικτική λειτουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εσείς αποφασίζετε, όχι ο οργανισμός. Ο οργανισμός σας υποστηρίζει με καλά δεδομένα και αναλύσεις για να μπορείτε εσείς να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και εδώ ε, υπάρχει μια παράλληλη πορεία με το έργο του οργανισμού ε, στο οποίο υπηρέτησα στον ΟΗΕ. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να σα αναφέρω και να σε ευστήσω την προσοχή ω προ τι ανάγκες και τι πρέπει να πληρεί ω προσόντα ο διευθυντής είναι το βιογραφικό του. Θα πρέπει να έχει αποδείξει ότι έχει εργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία σε στόχου υψηλού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπορούσα να σα δώσω πολλά παραδείγματα. Το πιο πρόσφατο, μόλις πέρυσι, υπήρξε μια μεγάλη πρωτοβουλία για να ενισχυθούν τα συστήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη και αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από ένα ε, έργο ε, που ήταν η διαδικασία του Δουβλίνου ε, όπου εγώ ηγήθηκα 80% των συστάσεων προήλθαν από εκεί, από την παγκόσμια διαβούλευση που είχα κάνει μια τριετία και κατέληξα σε 100 συμπεράσματα. Ε, θα πρέπει να αποδείξει λοιπόν κανείς ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο απαιτήσεων και στόχων του οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριο Φλάχερτη. Εδώ ολοκληρώνεται η εισαγωγή σας και προχωρούμε στις ερωτήσεις. Είναι και για μένα νέα διαδικασία, είστε ο πρώτος στη σειρά. Πρώτη ερώτηση για τρία λεπτά από την πρώτη συντονίστρια. Α, ένα λεπτό ερώτηση και δύο απάντηση. Η κυρία Μόνικα Χόλμα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Μόνικα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα αγγλικά. Okay. Please go ahead. Following commissioners... Μετά ε, τα όσα εξήγηλε ο κύριος Τίμερμανς, κλείνει το μικρόφωνο. Your microphone is now Again. On. Ε, δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Ανοχή λοιπόν και πώς ε, θα καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, την ισλαμοφοβία, τον αντιχριστιανισμό και διάφορες άλλες μυσαλλοδοξίες. Πώς μπορείτε εσείς να συνεισφέρετε σε αυτή τη συζήτηση. Μισό λεπτό να βάλω και το ρολόι, το χρονόμετρο. Thank you Ευχαριστώ. Νομίζω η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική και άκουσα και εγώ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς να λέει ότι θα ενισχύσει αυτό το πλαίσιο για τη λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς συμμορφούνται τα κράτη-μέλη. Ε, πολύ σωστά τα λέει. Το βασικό θέμα είναι τα εξή τρία. Στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί με διάφορους τρόπους εκεί να εμπλακεί. Πρώτον, όπως ήδη πράττει, να έχει αξιόπιστα στοιχεία για τα γεγονότα αυτά, το, το, τα εγκλήματα μίσου και τις ομιλίε μίσου, αυτέ τι κατηγορίες που ε, αναφέρονται. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα. Το είδατε στην απάντηση στην κατάσταση με το Σαρλί Εμπτό. Μπορεί να γίνει καλή δουλειά μέσα σε ένα μήνα και μόνο. Και τέτοια στοιχεία μπορούμε να έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο και αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεύτερον, ε, ο οργανισμός έχει ρόλο να παίξει για ε, τα τεχνικά, για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν συμφωνούν πάντα όλα τα κράτη-μέλη και πού τραβάς τη διαχωριστική γραμμή. Εκεί που λέει ο νόμο κατά τη γνώμη μου και ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να δίνει τεχνική και νομοτεχνική συμβουλή. Και αυτό ε, θα ευοδοθεί ω προσπάθεια το συμπόσιο που λέει ο κύριο Τίμερ μα, μόνο εάν τα αποτελέσματα διαδοθούν. Και εκεί έχουμε ρόλο να παίξουμε, Οργανισμό, δηλαδή σε επίπεδο κρατών μελών, γιατί εκεί πραγματικά θα ε, γίνει διαφορά. Ευχαριστώ. Και πάλι ένα λεπτό και ένα δίλεπτο απάντηση ο κύριος Νίτερ Μίλος, σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά όχι... Α, η Μάριου. Συγγνώμη, δεν σας διευκολύνω. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Μάριου Τόριστη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριο Φλάιρτ, έχετε εντυπωσιακό βιογραφικό. Έχετε ασχοληθεί με όλες τις σημαντικές στοιχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ξέρετε σε αυτή την Επιτροπή αναμένουμε ε, το FRA να είναι ένα σημαντικός μας εταίρος ε, συνεργάτης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχετε ένα ολοκληρωμένο μέσο ώστε να συγκρίνεται τα κράτη-μέλη και να διαπιστώνεται κατά πόσο τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σήμερα είχαμε μια έκθεση ε, του FRA, αλλά δεν ήταν ε, αυτή η καθολική ευκαιρία να έχουμε δηλαδή δείκτες συγκρίσιμους για όλες τις χώρες. Εσείς πώς τα βλέπετε, είναι μια ρεαλιστική προσδοκία, θα μπορέσει το FRA υπό τη δική σας διεύθυνση να το ολοκληρώσει αυτό, δηλαδή να μας δώσει αναχώρα ε, εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λόριστον ήμουν παρόν στην ε, πρωινή έκθεση. Πιστεύω πως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωματών ακολουθεί την επιθυμητή από εσά κατεύθυνση. Ε, δεν μιλά αφηρημένα για προβλήματα, ε, μιλά για το πού υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά και μιλά και για καλή πρακτική, πολύ σημαντική λειτουργία. Οι δείκτες και η μεθοδολογία που ακολουθεί ο οργανισμός και έχει προτείνει και εφαρμόζει σε όπως η Ρωμά ας πούμε, ή τα παιδικά δικαιώματα είναι ε, η συγκέντρωση των στοιχείων ε, σε τέτοιο επίπεδο όπως αυτό που χρειάζεστε για να κάνετε χρήσιμες συγκρίσεις. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε αυτό να το καταφέρουμε. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε υπόψη ότι Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνέστησε την FRA ως οργανισμό εποπτείας την συνέστηση ώστε να σας δίνει πραγματικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πως αυτό μπορεί να ενισχυθεί, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι επίσης προχωρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο ερώτημα από την κυρία Helga Stevens από την ομάδα ECR. Ένα λεπτό για την ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα και εγώ την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Κοίταξα και την έκθεση, την ετήσια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και υπάρχει ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο ε, για τα άτομα με αναπηρίες και γίνεται και παραπομπή στη σύμβαση του ΟΗΕ που είναι η μόνη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω για τα άτομα με αναπηρία που έχει κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε κι εσείς, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, είναι ένα κέντρο αριστείας και θέλει ε, ως ε, τέτοιο κέντρο να προβληθεί. Εσείς λοιπόν πώς το βλέπετε αυτό το κέντρο αριστείας, πώς βλέπετε το ρόλο του και την εφαρμογή της σύμβασης για τα άτομα με αναπηρία, συγκεκριμένα δηλαδή. Πώς το φαντάζεστε. Και αυτό το mainstreaming, δηλαδή η ένταξη αυτών των θεμάτων σε όλες τις πολιτικές και για τα άτομα με αναπηρίες. Κάτι που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πολύ συχνά υπάρχουν διακρίσεις και η κάθε κατηγορία ε, εξετάζεται χωριστά. Ε, έχουμε ανθρώπους ε, ε, που είναι άτομα με αναπηρίε ή που μπορεί να είναι ε, ομοφιλόφιλοι ή που μπορεί να είναι ξένοι μετανάστες και καμιά φορά έχεις μία μαύρη που μπορεί να είναι ανάπηρη και ομοφιλόφιλη. Τι γίνεται με Ναι, έχουμε την, συνυπογράψει την ε, σύμβαση για τις ε, αναπηρίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, στην ουσία είναι υπόλογη για κάθε παράβαση σχετικά. Πάντως η Ευρώπη ήδη έχει θεσπίσει πολύ υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και δίνει το καλύτερες πρακτικές. Επίσης έχουμε και στοιχεία κλειδιά για το πώς εφαρμόζονται οι καλύτερες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι λογική, το λογικό κατάλημα. Σε ποιο βαθμό αυτό αντιμετωπίζεται στα κράτη-μέλη και από τα ίδια τα θεσμικά όργανα. Και δεύτερον, εξαιρετικά, δεύτερη πρόκληση είναι το θέμα της ε, χορτικότητας πώς το υποκείμενο αυτό γίνεται σεβαστό ακόμα και όταν ζει με κάποια αναπηρία. Εμείς λοιπόν συγκεντρώνουμε στοιχεία ώστε να μπορέσετε εσείς να καταλήξετε σε συμπεράσματα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Στίβεν σε σχέση με αυτό που λέμε στα θεμελιώδη δικαιώματα, την διατομιακότητα του αναπηρία. Όταν δηλαδή κάποιος ε, υποφέρει από κάποια αναπηρία και ταυτόχρονα τυχαίνει να είναι και στην ομάδα των ε, LGBT ή e, να προέρχεται από κάποια μειονότητα ε, όπως η Ρωμά, σίγουρα θα έχει ε, ακόμα μεγαλύτερο αρνητική εμπειρία. Η ανάλυση λοιπόν της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι διατομεακή, να αναγνωρίζει την περιπλοκότητα της ταυτότητάς μας και του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά στοιχεία του χαρακτήρα μας και της προέλευσής μας ε, μας ε, αλληλεπιδρούν και μας κάνουν να υποφέρουμε περισσότερο λιγότερο από το γείτονά μας. Ευχαριστώ. Μονόλεπτη ερώτηση Σόγκορ από το ΕΛΚ. Διακόπτει ναι, ο ζητώ συγγνώμη. Λάθος έκανα. Γιατί η επόμενη ερώτηση πρέπει να προέλθει από τη Σεσίλια Βίξτρομ, από την ομάδα Άλτε. Ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη και από τον υποψήφιο, η Σεσίλια Βίξτρομ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Φλάρτη, οι πανεπιστημιακές σας, ε, τα πανεπιστημιακά σας προσόντα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, οπότε δεν θα σας κάνω ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Τώρα, ε, ο μελλοντικό διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι και καλός διαχειριστής. Θα ήθελα λοιπόν, ε, αν μπορείτε, να μας πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό. Έχετε εμπειρία από τη διαχείριση κάποιου οργανισμού μεγέθους παρομοίου με την ΕΦΑΡΕ, πώς ε, πόσα άτομα είχατε υπό την διαχείρισή σας, ποιον προπολογισμό είχατε και ήσασταν υπεύθυνο γι' αυτόν και για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι και πιο προσωπικοί. Ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ενός, ε, μιας υπόθεσης ενός προβλήματος διοικητικού ή διαχειριστικού, το οποίο χειριστήκατε ε, στο παρελθόν και ήσασταν επιτυχής. Και τα πήγατε και πολύ καλά με τον χρόνο μου. Ναι, πολύ καλύτερα από μένα σίγουρα, λέει ο πρόεδρο. Και πάλι το συγγνώμη που τον εσά, κύριε υποψήφι, έχετε δύο λεπτά. εδώ τώρα δεν ξέρω αν εγώ θα είμαι ε, στην ώρα μου για να απαντήσω. Ναι, έχω διαχειριστεί οργανισμού εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Έχω διαχειριστεί τι επιχειρήσει επιτόπου το ε, ε, ε, σειράξει στη Βοσνία πριν από 20 χρόνια και πιο πρόσφατα σε μέρη όπως η Σιάρα Λεόνε, εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες επιχειρήσεις ε, ε, εν μέσω πολέμου. Είχαμε σε μεγάλες ομάδες και σημαντικό προϋπολογισμό όταν ήμουν συντονιστής των προγραμμάτων για την Ασία και τον Ειρηνικό στο τη Αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όταν πρόκειται για το προσωπικό είχα υπό την ε, διεύθυνσή μου 200 ανθρώπου. Δεν θυμάμαι όμω τον προπολογισμό ακριβώς, οπότε καλύτερα να μην αναφερθώ σε στοιχεία. Πιο πρόσφατα ε, εγώ διαχειρίστηκα την ε, Επιτροπή της Βόρειας Ιρλανδίας. Πολύ μικρή επιτροπή, ήμασταν 20-30 άνθρωποι, αλλά ασχολούμασταν με ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως οι, δημόσιο, οι περικοπές στο δημόσιο προπολογισμό και σε πολύ δύσκολο πλαίσιο. Και αυτό αφορούσε την επιτυχή μείωση μιας επιχείρησης που μέσω της περικοπής του προπολογισμού, πράγμα που δεν οφειλόταν στην ίδια την Επιτροπή, ε, ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί χρειάστηκε να, να το πλοίο στην πορεία του, ενώ λειτουργούσαμε με πολύ λιγότερους πόρους και έπρεπε να διώξουμε κόσμο. Ε, βεβαίως λυπήθηκα πολύ για τον ανθρώπινη πτυχή αυτής της υπόθεσης, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω ότι ήταν επιτυχής.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 Ε, θα πρέπει εσείς τώρα να πάρετε το λόγο και να θέσετε την ερώτησή σας στον υποψήφιο. Ένα λεπτό έχετε. Η ερώτηση από τους Πρασίνους, η σε Αρζεντίνη. Κύριε Φλάτη, είπατε μόλις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, συνέστησε την ω ως ε, σώμα εποπτείας, ως οργανισμό εποπτείας. Και ακριβώς είναι και εκεί, εκεί και η δυσκολία, γιατί πολλοί από εμά στο Κοινοβούλιο θα θέλαμε να παίξει και εποπτικό ρόλο ο οργανισμός αυτός. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι, όπου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, ορόσημα που να συγκρίνουν τη μία χώρα με την άλλη, όπου παίζονται παιχνίδια για τη χρηματοδότησή σας και τον ετήσιό σας και προσχεδιασμό, πρόγραμμα εργασίας και την επιθυμία μας ε, για σύνταξη ε, νομοθεσίας σχετικής με τα θεμελιώδη δικαιώματα που βασίζεται στα, δικά, στα στοιχεία που εσείς συγκεντρώνετε. Πώς βλέπετε λοιπόν τον πολιτικό ρόλο του οργανισμού αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαργεντίνη. Ο ρόλος του οργανισμού είναι να δίνει ε, τις πληροφορίες που χρειάζονται οργανισμοί όπως οι θεσμικά όργανα όπως τα δικά σας για να προβούν στη λήψη αποφάσεων. Φυσικά αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι άμεμπτα και να δίνουν ε, τις πληροφορίες που, για το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκρίσιμα με το διεθνή στάνταρ και το διεθνή χάρτη. Όμως το οργανισμό δεν μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ούτε κράτο μέλο. Αυτό θα ε, σήμαινε ότι θα έμπαινε στα χωράφια του Κοινοβουλίου των άλλων θεσμικών οργάνων. Εξεκολουθώ με είμαι τη ότι ο ρόλος του οργανισμού αυτού είναι υποστηρικτικός για εσά, για το πώ θα μπορέσετε εσεί να ενισχύσετε τα πλαίσια λογοδοσία. Και όπω το κάνετε αυτό, και γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το οργανισμό μα μπορεί να σα δώσει ειδική τεχνική αρρωγή. Ποια είναι τα διάφορα μοντέλα, πώ λειτουργούν στην πράξη, πώ μπορεί κανεί να επιστήσει την προσοχή στην ε, ε, χρηματοδότηση των υπαρχών των εποπτικών μοντέλων στην Ευρώπη. Πώς μπορεί κανείς να συνεργαστεί και όχι να ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα συστήματα του Συμβουλίου του Ευρώπης. Εκεί θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο. Πάντως η εποπτεία και το να δώσουμε κάποιο νόημα στα πορίσματά μας δεν είναι δικός μας ρόλος, έτσι όπως τουλάχιστον έχει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός. 11 ερωτήσεις από τα μέλη, λέει, μετά από την εισήγηση. Τώρα έχω το EFTD. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από το EFTD σήμερα εδώ? Όχι. Απλώς ρητορική το η ερώτηση. Έπρεπε να με ξέρετε μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, δεν έχουμε εδώ συνάδελφο από το e FTD. Ε, μειώνονται οι τάξεις είναι πέμπτη απόγευμα, πάντως θα συνεχίσουμε, αλλά ίσως είναι άδικο κάποιοι ε, συνάδελφοι να έχουν λιγότερες ερωτήσεις από ό,τι άλλοι. Θα πάμε στο τέλος και θα δούμε αν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να δώσουν μια ερώτηση, γιατί νομίζω πως είναι δίκαιο όλοι να έχει θέσει την ίδια αριθμό ερωτήσεων. Υπάρχει κανείς από το ΙΕΝΕΦ εδώ. Είναι μια νέα ομάδα. Ναι. Μόλις έφυγε. Ε, είναι ενοχλητικό, εν πάση περιπτώσει, Μόλι έφυγε. Μία εγγεγραμμένη, κανεί. Λοιπόν, τώρα κύριε Σόγκα, τώρα ήρθε η ώρα σα. Είστε αριθμό 10 από του 11, ζητώ συγγνώμη για προηγουμένω. Είσαστε από το ΕΛΚ, 10. Ευχαριστώ. Προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ε, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με παραδοσιακές εθνικές μειονότητες που υφίστανται ε, πολλά δεινά για τους γλωσσικούς νόμους, ε, για νόμους συλλογική ενοχής που ακόμα επικρατούν στην Ευρώπη. Πολλές περιπτώσεις ακούμε και από τον οργανισμό και από την Επιτροπή και τον ίδιο τον κύριο Τίμερμανς α, ότι αυτό είναι εθνικό θέμα. Ε, δεν είμαστε καλύτεροι μαθητές όλοι, αλλά η Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία, Σλοβακία, φέρω μερικού, είναι ορισμένα παραδείγματα. Ευχαριστώ κύριε Σόγκορ. Η πιο χρήσιμη απάντηση είναι να θυμίσω τον δυνητικό ρόλο που έχει ο οργανισμός να δώσει σάρκα και οστά και πνοή στο χάρτη σε εθνικό επίπεδο. Μερικές περιπτώσεις έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Μόνο 14% του πληθυσμού γνωρίζει το χάρτη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να το κάνουμε συνταγματικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη για να μπορούν οι εθνικοί φορείς να βασίζονται. Ο χάρτης έχει ε, πολλά να πει για τα δεινά πολλών μειονοτήτων, πολλών κατηγοριών και θα μπορέσει να χειραφετήσει πολλούς ενδιαφερομένους και θα έχει ευεργετική επίδραση στον τομέα που μόλις αναφέρατε. Άννα Γκόμες ήταν η ενδεκάτη και τελευταία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάλι για τον ρόλο, το ελεκτικό παρακολούθηση ή θα μπορούσε ο οργανισμός να βοηθάει τους ευρωβουλευτές δίνοντας στοιχεία αντίστοιχα με του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, που παρακολουθεί τον προϋπολογισμό. Εσείς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι αντίστοιχο για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Βλέπε τρόικα τα όσα συνέβησαν και ακόμα συμβαίνουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Δύο λεπτά παρακάτω. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Πάρα πολύ σύντομη απάντηση είναι ναι, καταφατική. Νομίζω ότι ο Οργανισμός Θεμελιδών Δικαιωμάτων θα καλωσόριζε περισσότερα αιτήματα ενημέρωσης για να υπάρχει αυτή η παραδοχή και η απόδειξη ότι είναι εγκάρσια η εφαρμογή παντού και υπάρχουν και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Βεβαίως ξέρω ότι υπάρχουν πολιετή πλαίσια λοιπά, Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι διακριτό, ξεχωριστό. Παρακολουθεί κάθε ε, πτυχή ε, της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και φυσικά είναι πολύ οικοδομητική ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Um, Ο Πρόεδρος Μωράης, έχω τώρα την εξής ιδέα θέσαμε ερωτήσεις στον υποψήφιο, έχει κάνει και την εισαγωγική του τοποθέτηση. Ε, περνούν τα περνία η ώρα. Πεστε μου λοιπόν, για να είμαστε έντιμοι και απέναντι στους άλλους υποψηφίους, γιατί είναι σημαντική η θέση αυτή και βεβαίως πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, ίσως βοηθήσει εάν αναλάβετε την δέσμευση να παραμείνετε ώστε να είναι ακριβώς η ίδια μεταχείριση και για τους τρεις υποψηφίους. Ήταν πραγματικά εξαιρετικές ερωτήσεις και καλύψαν μεγάλο έδαφος για να εξασφαλίζεται και η πολιτική ισορροπία. Συμφωνείτε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και τις επόμενες δύο υποψήφιες. Ορίστε. Η κυρία Βίκστρομ. Α, όχι, πρώτα η Τζούντι. Βεβαίω, ε, τον ίδιο αριθμό ερωτήσεων, αλλά όχι τι ίδιε ερωτήσει. Είναι τρία διαφορετικά άτομα, έτσι είναι. Ναι, ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε τι ερωτήσει, απαντά ο πρόεδρο Μωράη. Αλλά καλύψτε περίπου το ίδιο έδαφο, ε. η ίδια ποιότητα ερωτήσεων από τα ίδια πρόσωπα. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άλλε ερωτήσει δεν έχουμε για την ώρα για τον παρόντα υποψήφιο. Ορθών. Ωραία. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Ο Φλάχερτη. Ε, ζητώ συγγνώμη βέβαια για τα μικρά οριστήματα. Ευχαριστώ κύριε Φλάχερτη. Ας περάσουμε τώρα στην κυρία Βαντερλάν που είναι η επομένη υποψηφία. Καλώς ήρθατε κυρία Βαντελάν. Ορισμένοι σας γνωρίζουν, πρώην Ευρωβουλευτής. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν συμφωνείτε. Ο χρόνο είναι σχετικά περιορισμένο. Σα γνωρίζετε, είναι και πέντε απόγευμα. Είσαστε και πρώην Ευρωβουλευτή. Αντιλαμβάνεστε το ε, κάπω στενό τη ε, ε, καταστάσεως ε, να σας εξηγήσω πώς ε, θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ως υποψηφία καλείστε να τοποθετηθείτε για 5 λεπτά. Μετά από την εισαγωγή σας αυτή θα έχουμε ένα αριθμό ερωτήσεων από τα μέλη. Ανά ένα λεπτό για τον ή την ευρωβουλευτή για να υποβάλει την ερώτηση και δύο, μέχρι δύο λεπτά για την απάντησή σας και θα σας υπενθυμίζω ε, την πάροδο του χρονικού όριου. Θα είμαστε ήρωα στην τήρηση του χρονικού όριου, έτσι ώστε να είναι δίκαιη η μεταχείριση και των ε, τριών υποψηφίων. Βεβαίω μπορείτε να μιλήσετε όποια επίσημη γλώσσα επιθυμείτε και βεβαίω θυμίστε ότι μεταφράζεστε και μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Τοποθετηθείτε λοιπόν για πέντε λεπτά και μετά θα σας υποβάλλουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ κοντά σας. Ήμουν και αντιπρόεδρος της Επιτροπής σας επί δεκαετία. Μετά από την επίθεση στους διπλούς πύργους και η δική μας Επιτροπή κρίθηκε τότε να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις νέες ανάγκες. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Βεβαίω έχει τεθεί σε ισχύ και ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων προπενταετία. Και βλέπω, χωρίς να με εκπλήσει αυτό, ότι παραμένει η ε, κοινοβουλευτική σας επιτροπή ένα από τα θεμέλια. δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε πλήρη εξασφάλιση. Υπάρχουν υψηλά επίπεδα αντισημιτισμού, διακρίσεων σε βάρος αναπήρων, γυναικών, Ρωμά, ε, παιδιών, ρατσισμός, ε, κηρύγματα μίσους, διακρίσεις σε, βάση θρησκείας κλπ. Ο χάρτη είναι σημαντικό και θα χρειάζεται όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. όπω η Ευρώπη βρίσκει νέε απαντήσει σε σημαντικά προβλήματα οικονομικά και ασφάλεια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικέ που θα ασκούμε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, λαμβάνουν υπόψη τι ενδείξει για το τι πραγματικά λειτουργεί και ότι τέλο χρησιμοποιούμε του λίγους πόρου που διαθέτουμε σωστά. Και ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν ο, ο οργανισμός, ο FRA, να εξυπηρετεί εσάς. Γνωρίζω ότι είμαι διαφορετικού είδους υποψηφία, διότι για 8 χρόνια είχα και ερετό αξίωμα. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι πλεονέκτημα, διότι μου προσφέρει κάποιες ιδιότητες ε, που δεν έχουν άλλοι, γιατί έχω παρακολουθήσει συζητήσεις, ε, γνωρίζω πώς να επηρεάζω ε, μια ημερήσια διάταξη. Ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν ότι πρόκειται για ένα μειονέκτημα, διότι είχα μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Σε αυτού πάντω θα έλεγα εγώ ότι αντιλαμβάνομαι πλήρω ότι ο οργανισμό FRA μπορεί να είναι επιτυχημένο μόνο εφόσον είναι απολύτω ουδέτερο και παραμένει εντό των αρμοδιοτήτων του. Εγώ είμαι απόλυτα, ε, εγώ δεσμεύομαι απολύτω να το διατηρήσω αυτό. Όταν μπήκα ε, επικεφαλής του γραφείου του ανώτατου δικαστή στο ε, ποινικό δικαστήριο, ε, ακριβώς αυτό έπραξα. Ήμουν απόλυτα ουδέτερη. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένα όργανο βασισμένο σε συγκεκριμένε ενδείξει και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το αν θα στείλουμε τον κόσμο στη φυλακή ή όχι. Η πολιτική λοιπόν αφήνεται στα χέρια των πολιτικών. Αλλά πρέπει να του υπενθυμίζουμε το, τα, τα νομικά πλαίσια μέσα στα οποία οφείλουν να λειτουργούν. Και βεβαίω και οι δυνατότητε για να βελτιώνεται η απονομή τη δικαιοσύνη. Συμβατικές αποφάσεις λοιπόν, συμβατικές ανθρωπιστικές προκλήσεις όπως τώρα με τους πρόσφυγες και μετανάστες, ίσως να χρειάζεται να αποφασίσετε αν θα δώσετε νέους πόρου στη μάχη κατά του αντισημιτισμού ή των διακρίσεων. Κάθε φορά που θα διατυπώνετε τις πολιτικές αυτές, εγώ πολύ ευχαρίστως θα είμαι δίπλα σας για να σας προσφέρω τα δεδομένα βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα, σε πραγματικές ενδείξει. Ο οργανισμό FRA πρέπει να παραμείνει βασικός εταίρος της Ευρωβουλής. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να προωθήσουμε μια νοοτροπία βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η εμπειρία μου μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Στι συζητήσει που διεξάγονται και που συνεχίζουν να διεξάγονται στην συλλογή δεδομένων που θα τεθούν υπόψη σα ημών του ε, Συμβουλίου άλλων οργανισμών έτσι ώστε να επιτύχουμε maximum impact. Το όραμά μας και η στάτευσή μας είναι σημαντικά. Βεβαίως δεν είναι μόνο ο διευθυντή, αλλά είναι το διοικητικό συμβούλιο σε συνεργασία με του άλλου εταίρου αυτά που εγκρίνουν τι προτεραιότητε. Χρειάζεται βεβαίω και έναν έμπειρο μάνατζερ ο FRA για να επιβάλλει τι προτεραιότητε αυτέ και για την σωστή χρήση του προπολογισμού και την ε, στάτευση του προσωπικού. Εγώ είχα τις αρμοδιότητε αυτές για θέματα δημοσιονομικά, για 90 ε, ανθρώπους προσωπικό πλήρους απασχολήσεως στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στρατηγικός σχεδιασμός, ε, προϋπολογισμός και ούτε καθεξής. Το ICC έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 100 εκατομμυρίων και χίλια πρόσωπα προσωπικό. Εγώ είχα ιδρύσει και επιτροπές. Ο FRA θα είναι τόσο αποτελεσματικός όσο η δράση του προσωπικού του. Και εγώ ευχαρίστως θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία που διαθέτω για να το επιτύχω αυτό. Η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις και υπάρχει ο κίνδυνος τα ανθρώπινα δικαιώματα να θεωρηθούν είτε αυτονόητα είτε και μια πολυτέλεια. Όχι, πρέπει να είναι απόλυτα εγγυημένα. Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα που δαπανά ο FRA δαπανώνται για να βρεθούν πραγματικές μακροπρόθεσμες λύσεις. Εγώ θα θεωρήσω μεγάλη μου τιμή να μπορέσω να συμμετάσχω στην προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαντελάν. Ας προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στις ερωτήσεις και η πρώτη θα γίνει από την κυρία Μόνικα Χόλμαερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας παρακαλώ ερώτηση ενός λεπτού και απάντηση εντός διλέπτου. Κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μόνικα Χόλμαερ, ε, ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν και είναι σε πολλούς τομείς πραγματικά δραστήριος. Δραστηριοποιείται και σε τομείς όπου υπάρχουν ήδη εξειδικευμένοι οργανισμοί ή θεσμικά όργανα. Υπάρχουν λοιπόν οι πολυσμένε περιστάσει εκεί και επικαλύψεις και ανάγκη συνεννόηση με του άλλου αυτού τους οργανισμούς. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε στη συνεννόηση με άλλα συναρμόδια όργανα, οργανισμούς κλπ. ενδεχομένως να αποφύγετε την επικάλυψη ή να αποφύγετε να κάνετε μελέτες που κάνουν και άλλοι, πώς θα συνεργαστείτε με άλλους οργανισμούς που συνδέονται και θεματικά με τον FRA, πώς θα συντονιστείτε επί της ουσίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε και τα δεδομένα που ενδεχομένω προσφέρουν άλλοι οργανισμοί. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Έχει ναι, δύο λεπτά, έχετε το λόγο. Απαντά στα γερμανικά. Η υποψηφία, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα, για παράδειγμα το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ε, ε, αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ΩΣΑ κλπ. Ε, αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και δεν μπορούμε να επικαλυπτόμεθα. Βλέπουμε ήδη ότι η FRA ε, έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, για παράδειγμα με την ΑΣΟ τον Frontex κλπ. Και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει η συνεργασία αυτή. Για την Frontex έριξα πάλι μια ματιά, είπαμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τη στρατηγική για την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο έργο. Έχουμε και την ε, ε, ε, αστυνομική σχολή, την πολύ Academy. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στα μαθήματα της, πολιτικής ε, πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Πού μπορούμε να συνεργαστούμε δηλαδή με άλλους, πού μπορούμε να παίξουμε καλύτερα εμείς ένα ρόλο έτσι ώστε να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την, ε, τις θετικές επιπτώσεις του έργου μας. Έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε μια μονάδα, δεν συγχωρείτε. Ναι, έλεγα λοιπόν αυτή η συνεργασία κινείται καλά, νομίζω μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή θετική επίπτωση των δράσεών μας. Επόμενη ερώτηση. Κρίσνη Τεμίλερ από τους σοσιαλιστές. Ένα λεπτό έχετε. Δεδομένων των δυσκολιών που αυξάνονται διεργώ για τους Ρωμά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την παιδεία, τι διακρίσεις ε, στον τομέα της στέγασης, της υγείας αλλά και της αγοράς εργασίας, ποιος είναι ο στόχος σας ε, στην ε, μελλοντική σας συντολή όσον αφορά τις στρατηγικές ένταξεις των Ρωμά, ώστε να δοθεί νέα πνοή σε αυτές τις ε, εν λόγω στρατηγικές. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως οι περισσότεροι στόχοι έχουν περιγραφεί σε εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά. Αυτό που νομίζω όμως ε, είναι σημαντικό είναι όντως να εφαρμοστούν αυτές οι στρατηγικές όπως έχουν ε, ορίσει τα κρατημέλη και για να γίνει αυτό είναι φυσικά να παρακολουθούμε την κατάσταση και η Κομισιόν είναι σαφής ε, ότι υπάρχει ρόλος για το ΦΡΑ εδώ αλλά βέβαια πρέπει ακόμα να γίνει πολλή δουλειά. Στέγαση, παιδεία, απασχόληση. Οι διακρίσει ε, εξακολουθούν να υπάρχουν και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι Ρωμά θα μπορέσουν πλήρω να συμμετέχουν και να χαίρουν των θεμελιωδών του δικαιωμάτων. Ο ρόλος λοιπόν του ΦΡΑ είναι όχι να θεσπίσει νέους στόχους ή να τους αλλάξει αυτούς που υπάρχουν, αλλά να εργαστεί με τα κρατημέλη με τη βάση των υφιστάμενων στόχων για να επιτυχθούν δεν είναι εύκολο. Ε, και το νέο σχέδιο του ΦΡΑ είναι να δουλέψει σε τοπικό επίπεδο, να πάει δηλαδή στις τοπικές κοινότητες, να δει ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια που όχι μόνο αντιμετωπίζουν οι Ρωμά αλλά και οι μη Ρωμά. Και να δει μετά πώς και τι λειτουργεί επί τόπου. Να δούμε λοιπόν που έχουμε υποσχόμενα προγράμματα, που έχουν πραγματικά αποτελέσματα, πραγματικά επιτεύγματα και να δούμε που αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν μπορούμε χρόνο με το χρόνο να αναλύουμε τα στοιχεία και να εξακολουθούμε να λέμε η κατάσταση είναι ακόμα άσχημη και είναι ακόμα άσχημη. Πρέπει να πούμε τι λειτουργεί, ποιο πετυχαίνει κάτι και μετά να προσπαθούμε αυτό να το διαδώσουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι πώ οι πόροι θα, εφαρμο... θα χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ από την ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω και εγώ από πλευρά μου. Πώς φαντάζεστε την εφαρμογή του άρθρου 14 εδάφιο 4 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που δεν θέλουν να προβάλλεται στο σχολείο στα παιδιά τους στα μαθήματα η ομοφιλοφιλία ως κανονική συμπεριφορά. Σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σλοβακία και στην Κροατία έγιναν δημοψηφίσματα και οι γονείς μαζικά διατράνωσαν ε, την αίσθησή τους ε, και την άποψή τους και στη συνέχεια χώρες αυτές υπέστησαν επιθέσεις που έκαναν αυτά τα δημοψηφίσματα. Εσείς τι θέλετε να κάνετε για να προωθήσετε τα δικαιώματα των γονέων αυτών βάσει του άρθρου 14 εδάφιο 4 του χάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Το άρθρο 14 έχει να κάνει με το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Και παρόλο που υπάρχει σαφές δικαίωμα στην εκπαίδευση, δεν θα πει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τι θα διδάσκει κάθε σχολείο σε κάθε κράτο μέλο. ούτε ποιο θα είναι το πρόγραμμα σπουδών του κάθε σχολείου. Η διδακτέα ύλη. Αυτό νομίζω είναι υπερβολικό. Ετίθεται όμω ένα θέμα το οποίο θέσατε κι εσεί για του ΛΟΑΔ ε, που θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στα σχολεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που υπήρξε πρωτοπόρα και ήταν η πρώτη που επέτρεψε το γάμο μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών. Και τώρα ζω σε μια χώρα που είναι η Σλοβενία και ανοίγει σιγά σιγά αυτή η προσπάθεια. Τι βλέπω, νομοθεσία είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης, γιατί όταν έχεις ε, ισότητα στο νόμο δεν σημαίνει ότι ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής ή ότι οι μαθητές αισθάνονται άνετα στο σχολείο ή δεν μπορούν να εκδηλωθούν γιατί θα τους δίνουν ή θα έχουν άλλες βίες εκδηλώσεις και πραγματικά ε, το επίπεδο της βίας κατά τον ΛΟΑΔ στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει απαράδεκτα υψηλό. Το ίδιο νομίζω ισχύει και με τους Ρωμά. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω δεν είναι μόνο να παρακολουθούμε εμείς την κατάσταση και χρόνο με το χρόνο να αναφέρουμε ότι η κατάσταση είναι άσχημη και τον επόμενο χρόνο το ίδιο ή μπορεί να έχει επιδεινωθεί κιόλα, αυτό που θέλω να δω είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση στις κάτω χώρες, ε, ε, ε, στη χθινομοθεσία στην πατρίδα μου, έτσι ώστε να υπάρξει εκπαίδευση και θέλω να δω αν αυτό θα επιτύχει και αν επιτύχει να μοιραστούμε τις εμπειρίες και άλλα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ή τα Εθνικά Κοινοβούλια ή εσείς και εμείς έχουμε focal points, σε μία επαφή στα διάφορα κοινοβούλια για να γίνονται παντού σεβαστά και ε, ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των σεξουαλικών μειονοτήτων. Η Σεσίλια Βίξτρομ από τους φιλελευθέρους θα κάνει την επόμενη ερώτηση. Ένα λεπτό έχετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι ε, είχατε εμπειρία ως προσωπάρχης Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και είπατε ότι θα σας ε, χρησιμεύσει αυτή η εμπειρία. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια παραπάνω, πώς θα γίνει αυτό. Ε, τι ε, θα γίνει, γιατί αυτή η εμπειρία σας ήταν σε ένα δικαστήριο. Πώς θα μπορέσετε να την αξιοποιήσετε σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει και αντιστοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας είπα προηγουμένως ότι έχω εμπειρία στη διαχείριση του προσωπικού του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου ήταν πολύ διαφορετική μεταξύ του υπάλληλοι. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα σώμα δικαστικό που πρέπει να λειτουργήσει σε ένα πολιτικό κόσμο. Είχε ε, εκφραστεί μεγάλη κριτική και από την Αφρικανική Ένωση, γιατί αντιμετωπίζεται το Σουδάν και όχι τη Συρία. Αυτό δεν το επιλέγει το δικαστήριο, αλλά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμείς έχουμε μια εντολή και θα πρέπει στα πλαίσια της εντολής μας να δράσουμε. Αντίστοιχα είναι και ο οργανισμός ΦΡΑ, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολλοί θα ήθελαν να προχωρήσει περισσότερο, αλλά έχει μια εντολή και εντός αυτής πρέπει να κινείται. Αυτό είναι πολιτικός κόσμος. Έχουμε ανεξαρτησία, αλλά έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο και καλό είναι να ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό. Άλλο παράδειγμα. Είχαμε πολύ έντονη συζήτηση για την ειρήνη και την ε, δικαιοσύνη ή την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους. Είναι η ίδια ε, ούτε καν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι η ίδια όψη του, του νομίσματος. Και τέλος, στο μισό λεπτό που μου μένει, όταν πήγα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, 95% του προσωπικού ήταν, ήταν ποινικολόγοι, που εγώ δεν είμαι. Και το καλό είναι ότι φέρνεις νέες δεξιότητες. Ακριβώς εγώ ε, δεν είχα μια καριέρα 10 ετών στο ποινικό δίκαιο, είχα μια εξωτερική ματιά. Και ως διευθυντής του ΦΡΑ δεν θέλω να είμαι επικεφαλής επιστήμων και ευρύτρια ε, και βασεύομαι σέβομαι όλους τους ερευνητές, αλλά θέλω να ε, δανειστώ την εμπειρία και τη γνώση που έχουν και να μεγιστοποιήσω το όφελος που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή. Η κυρία Λούνατσεκ από πλευράς των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εγώ δεν ήμουν μέλος ε, όταν ήσασταν εσείς και χαίρομαι που σας γνωρίζω. Είπατε και ήδη ότι καμιά φορά, ιδιαίτερα σε καιρούς ε, οικονομικής δυσπραγίας, πολλοί θεωρούν τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα ως πολυέλεια. Πολυτέλεια, συγγνώμη. Ε, και σήμερα κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ο οργανισμός είναι παραβίαση κατά κάποιο τρόπο της επικουρικότητας και θέλουν να διατηρήσουν την ε, κυριαρχία τους για θέματα που μπορεί να φαίνονται συγκρουσιακά, δικαιώματα ΛΟΑΔ, ισότητα φύλων, δικαιώματα παιδιών, γυναικών κτλ. Τι θα κάνετε απέναντι σε αυτούς τους πολιτικούς ή τα κράτη-μέλη, πώς θα τους πείσετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ε, είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε επιτίθενται ή παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών. Κοιτάξτε, εύκολο είναι αυτό, γιατί όλοι έχουν υπογράψει το χάρτη, όλα τα κράτη-μέλη και τα εργαλεία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σύμβαση για τα άτομα με αναπηρίες, διάφορες συμβάσεις του ΟΗΕ, είναι συμβατικές υποχρεώσεις τους που τις έχουν κυρώσει με πλήρως δημοκρατικές διαδικασίες, με εθνικά κοινοβούλια κτλ. Δεν επιβάλλουμε τίποτα σε κανένα, ο καθένας επιλέγει ο καθένα επιλέγει να δεσμεύεται από τις συμβάσει που προσυπογράφει. Βέβαια η πραγματικότητα διαφέρει από τη θεωρία. Πάντα θα πρέπει ο καθένας να επιλέγει τα στοιχεία και τα γεγονότα που συνδέονται με αυτά. Όταν βλέπετε τα γεγονότα, αυτά σας καθοδηγούν αυτόματα δείχνουν τα προβλήματα, δείχνουν ποια κράτη-μέλη προχωρούν καλύτερα. Και θα πρέπει να συνεχίζουμε να συζητούμε, να πιέζουμε, να πείθουμε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο δουλειά δική μας. Τόσοι συνάδελφοι, ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, τα θρησκευτικέ οργανώσει είναι πάρα πολλοί φορεί στην Ευρώπη και αν συνεργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πίεση και δεν είναι καθόλου πολύ τέλεια. Και είναι βασική ευρωπαϊκή αρχή και αξία. Ευχαριστώ. Έχουμε τη νέα ομάδα ε, ε, ε, Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας και ήρθε η συνάδελφος από την ομάδα αυτή. Έχετε το λόγο, κύριε Μάγερ. Ευχαριστώ, κυρία Φαντρελάν. Πριν από λίγα χρόνια είπατε ότι υπάρχει ένας Ισλαμικός πυλώνας στην Ολλανδική κοινωνία. Ως διευθύντρια, τι θα κάνετε για τον πυλώνα τον Ισλαμικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλεί την Ευρώπη. Τι θα κάνετε για να καταπολεμήσετε αυτή την απειλή. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για κάθε ομάδα που δεν αισθάνεται καλά στην Ευρώπη, δεν αισθάνεται ότι ανήκει στην Ευρώπη ε, και δεν θεωρεί ότι εντάσσεται στην κοινωνία. Εγώ δεν θα κάνω εδώ καμία διάκριση ε, ανάλογα με την προέλευση ή τη θρησκευτική προέλευση. Όταν το είπα και συμφωνώ, κάναμε μια συζήτηση για την ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία, για την εστομάτωση και στην Ολλανδία και στην Ευρώπη. Ε, Έχουμε μια πολυμορφία. Ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του ανεξαρτήτως χρώματος σεξουαλικής προτίμησης, θρησκείας και προέλευσης. Και αυτό είναι και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ισχύουν για όλους. Είναι θεμελιώδη και ως ε, διευθύντρια, εάν με διορίσετε, θεωρώ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας ποια είναι τα δικαιώματα και ότι ε, εφαρμόζονται για όλους. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές. Γνωρίζουμε Νομίζω ότι θα υπάρξει και το συμπόσιο αυτό που επίκειται για τον αντισημιτισμό, την Ισλαμοφοβία, τη διάκριση βάσης σεξουαλικής προτίμηση. Είναι όλες αυτές διαφορές. Αλλά το έργο μας δεν είναι να βάλουμε προτεραιότητες. Αυτό το κάνετε εσείς στο πολιετές πρόγραμμα, αλλά για να φροντίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα του καθενός είναι εγγυημένα. Thank you. I think Mrs. indicated Νομίζω η κυρία Χόλμαγε θέλει να κάνει την ερώτηση που έκανε προηγουμένως ο κύριος Σόγκορ. Για ένα λεπτό. Μια δεύτερη ερώτηση λοιπόν που έχει να κάνει με το πιο ευαίσθητο δωμάτι ε, που έχουμε στην κοινωνία, την πιο ευαίσθητη ομάδα που είναι τα παιδιά μας. Όλο και περισσότερο βλέπουμε νέες δυνατότητες και από το διαδίκτυο και διευρύνεται ε, η ομότητα, η βία σεξουαλικής φύσεως κατά μικρών παιδιών. Ε, τα σεξουαλικά κακοποιημένα και βαριά κακοποιημένα παιδιά αυξάνονται σε αριθμό πάρα πολύ και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, αυτά τα δύσκολα θέματα της κωδικοποίηση, τη κρυπτογράφηση, στην αστυνομία, τα έχετε υπόψη σα, η προστασία των δεδομένων. καθένα, έχει το δικαίωμα να προστατεύει στο διαδίκτυο τα δεδομένα του. Από την άλλη υπάρχει και η ανάγκη να διώκονται οι εγκληματίε στο διαδίκτυο. Εσεί ω διευθύντρια σε αυτό το πολύ ευαίσθητο τομέα πώς βλέπετε η μεγαλύτερη προστασία των παιδιών και να αποτρέπονται τα εγκλήματα ή να βοηθάτε να αποκαλύπτονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την εκτίμησή σας ότι είναι από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα αυτά και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύουμε όσο μπορούμε τα παιδιά μας. Όπως είπατε, και ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να ακρίβει και να συγκαλύπτει και τα εγκλήματά του κατά των παιδιών. Είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση αυτή που γίνεται για την ιδιωτική ζωή, για την ε, αποθήκευση δεδομένων, για την προστασία δεδομένων. Ένα από τα πρώτα που θα κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τον επόπτη προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων και να πόκειται σε εσά, τα κοινοβούλια και τους συναδέλφους σας από τα εθνικά κοινοβούλια, ε, πώς θα δείτε αυτά τα ζητήματα. Ο οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές. Μπορεί να υπάρχουν χώρες με καλύτερες επιδόσεις για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των παιδιών. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εγγυήσει που υπάρχουν εφαρμόζονται. Πολλέ φορέ δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία, αλλά εφαρμογή τη κείμενη νομοθεσία. Και βεβαίω εμεί υπάρχουμε για να σα βοηθούμε, να σα υποστηρίζουμε με μελέτε, έρευνε, στοιχεία και τάσεις. Βλέπουμε αύξηση στην κακοποίηση και χρησιμοποίηση του διαδικτύου για να κρύβονται τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή το διαπιστώσουμε, σας το λέμε, για να δράσουν οι πολιτικοί. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε χρόνο να περιμένουμε 4-5 χρόνια να αναλύσουμε και να δράσουμε. Και τελευταία ερώτηση είναι το κυρίου Νίτερ Μούλερ στη θέση της Άννας Γκόμες. Όχι, ανάποδα. Άννα, όχι εσύ, ο, ο Πίτερ θα τα πει. Okay, thank you very much. sorry, Anna. <coughs> Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη, Άννα. Κυρία Βανλάν, στην παρούσα κατάσταση σε ορισμένε χώρε μέλη είναι σαφές ότι οι μηχανισμοί κράτους δικαίου δεν επαρκούν. Πώς βρίσκεται, πώς βρίσκεται την ιδέα να αρχίσει μια διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης του κράτους δικαίου στις χώρε αυτές και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πώς βλέπετε μια επιβολή ε, του μηχανισμού για να εξετάσει την ε, τήρηση των κριτηρίων της Κοπενχάγης και μετά την ένταξη. Η υποψηφία. Σας ευχαριστώ. Όταν ε, συμμετείχα στο προσωπικό γραφείο του Επιτρόπου Βάντεν Μπρουκ για την ένταξη των νέων χωρών τότε με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αυτό ήταν πραγματικά ένα κέριο θέμα και κάναμε τις αιτήσει αυτές αναλύσεις, βεβαίως η Κομισιόν τις έκανε μόνο για τις υποψήφιες χώρες. Η διαφορά ανάμεσα στην προειδοποίηση ε, που απευθύνεται στην χώρα και μετά η χρήση του βαρύτατου μέσου του άρθρου 7, βεβαίως ε, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία εδώ υπέρ ενός μηχανισμού ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νέο πλαίσιο για το θέμα αυτό και η πραγματική, το πραγματικό θέμα είναι θα υπάρχει πολιτική συνένεση ε, για να ξεκινήσει κάτι το νέο. Αυτό βέβαια δεν είναι υπόθεση του Διευθυντού της Διευθυντρίας της FRA. Αν αποφασίσουν οι χώρες μέλη να το επεκτείνουν, τότε θα πρέπει η FRA να είναι έτοιμη να το πράξει, βέβαια εφόσον έχει τους απαραίτητους πόρους. Ταυτόχρονα υπάρχει τεράστιο ποσό πληροφοριών και μπορεί σχεδόν να πάρει κανείς και να αντιγράψει τις εκθέσεις που υπάρχουν για να κάνει έκθεση για τη συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, για ε, εγκλήματα μίσους, ας πούμε για τη Σλοβενία. Μπορείτε να τα βρείτε αμέσως όλες αυτές τις εκθέσεις και να τα στείλετε στους συναδέλφους σας και να δουν τι πρέπει να γίνει. Αν πάρετε λοιπόν τις εκθέσεις αναχώρα, τα διάφορα δεδομένα στις ειδικές εκθέσεις του, της, του οργανισμού FRA. Υπάρχουν ήδη από αυτά τόσα πολλά δεδομένα που μπορούν να μας επιτρέψουν να λάβουμε αποφάσεις. Αν αποφασίσετε να ιδρυθεί ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, τότε βεβαίω ο οργανισμό FRA θα είναι έτοιμο να συνεργαστεί μαζί σα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάντερλαν. Ευχαριστούμε για τι απαντήσει σα και για τη συμμετοχή σα στην ακρόαση. Σα ευχαριστώ και εσά κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, για τι ερωτήσει που θέσατε στην κυρία Βαν Ντερ Λαν. Uh, Μπορούμε να καλωσορίσουμε τώρα την κυρία Μπραντς και Χρύς. Βλέπω ότι πλησιάζει. Um, ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας και την επιμονή σας που παραμένετε μέχρι αυτή την ε, προχωρημένη ώρα. βεβαίω ευχαριστώ και το προσωπικό και όλες και όλους που έχουν παραμείνει μέχρι αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε κυρία Μπραντ και Χρύς. Είστε έτοιμοι? Α, τι ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λίγες ε, τώρα ε, ενδείξεις σχετικά με την διάρθρωση της διαδικασίας. Ως υποψηφία θα κληθείτε να προβείτε ε, σε πεντάλεπτη αρχική τοποθέτηση. Κάθετε λίγο μακρύτερα μου και καλά κάνετε. Θα σας εξηγήσω λοιπόν ότι πρώτα θα κάνετε μια τοποθέτηση των 5 λεπτών. Μετά θα σας τεθούν ερωτήσεις από τα μέλη μας σε χρονοθυρίδες των 3 λεπτών. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση. Θα είμαστε βέβαια αυστηροί με την τήρηση του χρονικού ορίου. Παρακαλώ μην υπερβείτε τα όρια αυτά. Υπάρχουν οι διερμηνείς, άρα μπορείτε να μιλήσετε όποια γλώσσα επιθυμείτε, αλλά παρακαλείστε όχι πολύ γρήγορα για να προλαβαίνουμε να σας μεταφράζουμε. Έχει το λόγο τώρα για τα πέντε λεπτά σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και είμαι ευτυχής που επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή. Θέλω να κάνω ε, κάποιες παρατηρήσεις στην εισήγηση αυτή. Η, μία, η πρώτη αφορά το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα όραμα για το πώς θα μετατραπούν οι αρχές ή ε, μάλλον οι, εικόν, οι απόψεις της Ένωσης σε συγκεκριμένες αρχές που καθορίζουν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. θέσπιση αυτού του οργανισμού το 2007 εξέφρασε μια δέσμευση ε, όλα αυτά να μετατραπούν σε μια επιχειρησιακή πραγματικότητα και ο οργανισμός αυτός είναι καινοτόμος οργανισμός για διάφορους λόγους έφερε, συγκέντρωσε μάλλον τα διαφορετικά, τους διαφορετικούς λόγους ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε μια κοινή προσέγγιση. Ε, υιοθέτησε μια πολύ ε, ε, διεπιστημονική μάλλον προσέγγιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, παρακολουθεί την συμμόρφωση ή παραβίαση βουλβάς των μελών των θεμελιώδων δικαιωμάτων, βοηθά τους οργανισμούς στη διατύπωση ε, πολιτικών με, επί τη βάση ε, στοιχείων που συγκεντρώνει και αναλύει ο οργανισμός καθώς και αναπτύσσει την μεθοδολογία ώστε όλα αυτά να καταστούν δυνατά. Τώρα, η αποτελεσματικότητα βεβαίως συνδέεται και με την εστίαση σε θέματα προτεραιότητας μέσα στο πλαίσιο του πολιετές βέβαια, του, μάλλον του πολιετούς ε, πλαισίου. Και επίσης ε, μπορούμε να δούμε ότι με βάση τα θέματα που σας απασχόλησαν πρόσφατα, το ΦΡΑ εστιάζει τις προτεραιότητές του στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων που έχουμε για τα πολύ επίγοντα ζητήματα όπως πρόσφατα με τη μετανάστευση, αλλά και με το θέμα της ε, παράνομης μετανάστευσης, την ρατσισμό αλλά και τα εγκλήματα βίας κατά εθνοτικών μειονοτήτων, LGBT και άλλων ευάλωτων μειονοτήτων. Πέρα από όλα αυτά το θέμα είναι μακροπρόθεσμο και επίσης εστιάζει ε, στην ε, εργασία κατά των διακρίσεων ε, για οποιοδήποτε λόγο εστιάζει στα δικαιώματα του παιδιού, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αλλού πρέπει να ανταποκριθούμε ε, χωρίς να αντιδρούμε όμως. Έχουμε την ευθύνη αλλά και την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη ώστε δραστήρια να εντοπίζουμε τα κενά στις πολιτικές και τα μειονεκτήματα ή τα προβλήματα μάλλον στην εφαρμογή συμβάλλοντας στην συνειδητοποίηση αλλά και στη θέσπιση θεματολογίου το mainstreaming των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών όπου τονίζονται σωστά τα θεμελιώδη δικαιώματα ως ε, κύριο σημείο προς παρατήρηση. Το ΦΡΑ βεβαίως ε, είναι προφανής ε, μέτοχος όλα σε αυτές τις εξελίξεις γιατί δίνει την εμπειρογνωμοσύνη του αλλά και στοιχεία αλλά και βασίζεται στη γενικότερη εικόνα για τη συνοχή και την καθολικότητα αυτής της διαδικασίας. Επίσης πρέπει να δούμε ε, πώς όλα αυτά είναι σχετικά, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε συνεργασία με όλους τους ε, φορείς κλειδιά ε, επιτόπου, ακούγοντας αλλά και παρέχοντας συμβολή και εμπειρογνωμοσύνη ως σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανεξάρτητα όργανα και βέβαια και στην κοινωνία των πολιτών, αν θέλετε, πέρα από τη ΜΚΟ, τον πανεπιστημιακό κόσμο και τους επαγγελματικούς οργανισμούς. Θα πρέπει να υπάρχει δραστήρια συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, με το Σύμβολο της Ευρώπης, κατεξοχήν συνεργάτης, καθώς και με το ΝΟΑΣΕ, και εννοώ συνεργασία όχι μόνο στα λόγια και στις ε, διακηρύξεις, όχι απλά δηλαδή να συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις, αλλά να διαβουλευόμαστε ε, στρατηγικά για να στοχεύουμε στη συνεργασία. Αυτή η φάση είναι μια φάση αλλαγής κατά εν ε, με πολλούς τρόπους, αλλαγές, καθώς έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα επιτροπή, αλλά υπάρχουν και επίγουσες ανάγκες γιατί Α, συγγνώμη, αλλά έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας και πρέπει να σας διακόψω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση για ένα λεπτό από το ΕΛΚΑ, η κυρία Χολμάγερ. Μόνικα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δημιουργήσει ένα συνεκτικό ε, νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να μπορεί να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και σχετικές διακρίσεις ή θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά παράθυρα στην νομοθεσία αυτή και αν ναι ως διευθύντρια θα ασχοληθείτε περισσότερο με την ε, εφαρμογή των διατάξεων αυτών περισσότερο ώστε να αντιληφθούν οι πολίτες μας στην καθημερινή τη ζωή ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και ποιου είδους δράσεις θα προτιμήσετε να αναλάβετε προς την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, απάντηση ω δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ αγαπητή κυρία Χόλμαϊερ. Νομίζω ότι όντω μπορούμε να είμαστε υπερήφανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που βασίζεται και όλα στο γεγονός ότι υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αλλά βέβαια και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το παράγωγο δίκαιο που προβλέπει αντιμετώπιση των διακρίσεων. Όμως, όπως έχουμε δει, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην εφαρμογή των υφισταμένων οδηγιών. Ένα από τα κενά στα οποία αναφερθήκατε στα παράθυρα είναι ότι χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος μέχρι ότου εγκριθεί η οριζόντια οδηγία. Συζητήσεις που διεξάγονται επίσης στα Εθνικά Κοινοβούλια για να προχωρήσει η ενίσχυση ε, του πλαισίου αυτού. Για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εδώ προβλέπεται ένας διτός ρόλος κατά τη γνώμη μου. Ασφαλώς ειδική στόχευση στην εφαρμογή και Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο, αλλά το πλαίσιο αυτό δεν μεταφράζεται σε πραγματική προστασία επιτόπου και ιδίω των πιο ευάλωτων προσώπων, που συχνά δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματα που διαθέτουν, ούτε με ποιον τρόπο μπορούν να τα προασπιστούν αποτελεσματικά ή ε, να προσφύγουν εφόσον αυτά παραβιάζονται. Εκεί ακριβώς πρέπει να στοχεύσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να προσφέρει δηλαδή, να συλλέξει δεδομένα, να προσφέρει τα απαραίτητα, τις απαραίτητες ενδείξεις και αποδείξεις και να προσφέρει την προστιθέμενη αξία με δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν πριν, κάνοντας έρευνες, συλλέγοντας τις υφιστάμενες πληροφορίες. Η Birgit τώρα από τους Σοσιαλιστάς και Δημοκράτας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση περισσότερο ε, στον χώρο της ομοφιλοφο... ομοφιλοφοβίας. Εκτός από τις προσπάθειες της Επιτρόπου, το, Συμβούλιο, το, ε, το Ευρωκοινοβούλιο κατά επανάληψη έχει ζητήσει και θεωρούμε ακόμα δυστυχώς ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση βλέποντας τον μεγάλο αριθμό διακρίσεων αλλά και βίων επιθέσεων κατά μελών της ομάδας αυτής. Μια στρατηγική υπέρ των διαφόρων ειδών ομοφιλοφίλων πώς θα έπρεπε να είναι και με ποιο τρόπο θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τη γνώμη σας. Μάλιστα, δύο λεπτά για να απαντήσετε, έως δύο λεπτά. Μάλιστα, η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, είναι σημαντικό θέμα. Μεγάλο και σημαντικό θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω έχει έρθει πια η στιγμή που βλέπουμε ότι ε, υπάρχει κάποια κίνηση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής όπως βλέπουμε και σε ορισμένες άλλες χώρες. Ασφαλώς δράσεις πολιτικής πρέπει να αναλυθούν. Όμως δεν είναι αυτός ο ρόλος ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει ήδη προσφέρει δεδομένα σημαντικά και σοβαρά που δείχνουν πραγματική αύξηση και αυτών που ακούμε από ομάδες θυμάτων και από οργανισμούς ή ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το νομικό πλαίσιο δεν είναι ε, πλήρες ταυτόχρονα βλέπουμε και τις εμπειρίες ε, εγκλημάτων μίσους και κηρυγμάτων μίσους. Εκεί, ωστόσο, στην προσπάθεια αντιμετωπίσης τους, δηλαδή έχει συμβάλει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και εξακολουθεί να ε, συμβάλλει, δείχνοντας ποια είναι η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής και επιτρέποντας την ε, άσκηση πολιτικών βασισμένων στις, στα δεδομένα που συλλέγει. Έχουμε και σε Προηγούμενε ερωτήσει που έχουν σχέση με τον διπλό ρόλο του FRA που αναφέρεται στην ανάλυση πιο συγκεκριμένα των ελλείψεων του ίδιου του πλαισίου ίση μεταχείρισης και προστασία των ε, ανθρώπων ε, που ανήκουν στην ομάδα LGBT. Χρειάζεται λοιπόν η ε, χρήση των εργαλείων που θα προσφέρει και με και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω την ερώτηση που έκανα προηγουμένως. Αλλά εσείς φυσικά δεν ακούσατε την ερώτησή μου. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 14 εδάφιο 4 του χάρτη. Το δικαίωμα των γονέων Ε, το δικαίωμα των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Υπάρχουν γονείς που αντιτίθενται ε, στο να εντάσσεται το θέμα της ομοφιλοφιλίας στη διδακτέα ύλη του σχολείου. Το βλέπουμε αυτό, αυτό να συμβαίνει σε διάφορα κράτη-μέλη. Η Κροατία και η Σλοβακία έκαναν δημοψηφίσματα σχετικά ε, και οι κοινωνίες μαζικά αντιτάχθηκαν στο γεγονός αυτό της ένταξης του μαθήματος λοιπόν υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιλαμβάνονται έτσι την ευθύνη τους ε, τη γονική. Εσείς πώς φαντάζεστε να ε, επιβληθούν και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των γονέων αυτών. Δύο λεπτά για να απαντήσετε το πολύ. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις και όλες οι ιδέες στα πλαίσια της ελευθερίας ε, του λόγου στην Ευρώπη και της σκέψης και χρειάζεται και σοβαρός διάλογος. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε ότι παρά τις διαφωνίες υπάρχουν εξελίξεις όλα αυτά τα χρόνια. Όταν εξηγούμε στον κόσμο τα δικαιώματα παρά ε, την ισχυρή θέληση να συμμετέχουν οι γονείς και να ε, επιλέγουν την ε, ανατροφή και την εκπαίδευση που θα δώσουν τα παιδιά τους και τα δικαιώματα των παιδιών. Τα ζητήματα των ΛΟΑΔ είναι τμήμα των θεμελιωδών αρχών και ελευθεριών, ισότητα, ίση συμμετοχή όλων στην κοινωνία και των παιδιών. Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ανοιχτό και να δέχεται ε, και να αποδέχεται όλους και τις μειονότητες λοιπόν τις ίδιες. Για το ρόλο του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι πρέπει αν δεν του ζητηθεί να επέμβει και να λέει ε, ποιες νομοθεσίες θα πρέπει να ισχύουν, να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα. Εκεί μπορεί να συλλέγει στοιχεία ο Οργανισμός Θεμελιδών Δικαιωμάτων και το βλέπουμε και στα πλαίσια της πολύ σοβαρής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σε πολλά ή τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη-μέλη, η ιδιαίτερη κοινότητα των ΛΟΑΔ, αντιμετωπίζει παρενόχληση και βία. Ευχαριστώ. Η Σεσίλια Βίξτρομ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση του διορισμού του επομένου διευθυντή θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που εσείς συμμετείχατε δύο χρόνια και είχαμε και συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την απαλλαγή του οργανισμού και έγινε μεγάλη ε, ανταλλαγή αλληλογραφίας γιατί υπήρξαν αιτιάσει ότι είχατε δώσει κάποιες συμβάσεις σε ΜΚΟ ε, ανθρώπων που ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή αυτό το έχετε ζήσει, μπορείτε να μας πείτε πώς λύθηκε αυτό το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήσασταν και εσείς αρμόδια. Τι πιστεύετε για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του οργανισμού και έχετε βγάλει συμπεράσματα και διδάγματα από την εμπειρία σας αυτή που θα θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό ερώτημα γιατί μπαίνουμε σε ζητήματα διακυβέρνησης και management. Βεβαίω συνδέονται αυτά τα δύο. Όντως υπήρξαν ζητήματα και στη δική μου περίπτωση όπου ο οργανισμός στη Λετωνία που ήμουν τότε εγώ ε, διευθύντρια ε, κέρδισε μία σύμβαση ε, για τον ΦΡΑ. Ε, τότε οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από λίγα χρόνια ήταν ήδη διαφανείς από τότε, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, συμμορφούμενες προς τις απαιτήσεις. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν δήλωση υπόθεν έσχες και εξήγησαν πώς έχει η κατάσταση. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση το έπραξα κι εγώ. Τότε δεν είχα ουδεμία σχέση. Ουδεμία ούτε ε, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε με την υλοποίηση. Ε, όλα αυτά ανατέθηκαν σε κάποιον με τον οποίο δεν είχα καμία επαφή. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι κανόνες για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ο προφανώς αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου, να κάνει ερωτήσεις και να βλέπει ε, αν είναι ικανοποιητικέ οι απαντήσεις. Εγώ πιστεύω στη διακυβέρνηση μπορεί καμιά φορά να αισθανόμαστε κάποια απογοήτευση ή κάποια ματέωση για το χρόνο που χρειάζεται η εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων και των διατάξεων και των εργαλείων διακυβέρνησης που είναι χρονοβόρα, αλλά κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ θεμελιώδης και για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για έναν οργανισμό που είναι τόσο ευαίσθητος όπως ο Οργανισμός Θελιδών Δικαιωμάτων με πολλές διαφορετικές απόψεις και τα λοιπά. Θα πρέπει να είμαστε απολύτως διαφανείς για να αποφεύγονται όλα αυτά. Η κυρία Σαρχεντίνη από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ιδιαίτερα επειδή έχετε υπάρξει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΡΑ, συχνά θα έχετε σκεφτεί ε, τι θα έκανα εγώ διαφορετικά και πώς εμείς από το ΦΡΑ σχετιζόμαστε με το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχε διάφορες επιθυμίες. Θα θέλαμε ας πούμε, να έχουμε ε, εθνικές εκθέσεις και το ΦΡΑ να παρακολουθεί, να υποπτεύει. Μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη. Εγώ πάντως θα το ήθελα αυτό. Τα κράτη-μέλη μπορεί να μην είναι απόλυτα ευχαριστημένα από τη δουλειά δουλειά που κάνει το ΦΡΑΙ και να μπλοκάρουν όπως κάποια χρόνια πριν την ε, δουλειά του ΦΡΑ. Επ' αυτό το φως εσείς ως νέα διευθύντρια του ΦΡΑ, τι θα κάνατε ή τι δεν θα κάνατε. Πού βλέπετε να βρίσκεται η δική σας θέση σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Thank Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα ε, που ε, Ε, αφορά το διοικητικό όργανο του ΦΡΑ. Είναι ανεξάρτητο σώμα που κάνει έρευνες, αλλά δεν είναι οργανισμός που λαμβάνει πολιτικής φύσης αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι ε, αλλωνών ε, Άρα εμείς πρέπει να λειτουργούμε με βάση τις αρμοδιότητες που έχουμε. Βέβαια υπάρχει συζήτηση για τον δυνητικό ρόλο στην εποπτεία ε, συγκεκριμένων χωρών. Πάντως δεν νομίζω πως είναι δική μου θέση να έχω γνώμη ή να πιέσω αν αυτό θα πρέπει να προχωρήσει. Όχι. Πάντως Ο στόχος είναι να, έχουμε συγκρίσιμα, να, να εκπονούμε συγκρίσιμα στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία από όλα τα κατημέλη συλλέγονται και ε, παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο. Εμείς έχουμε φόκ, ε, αιτία την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοιτάμε το σεβασμό των, των δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες. Τώρα, κατά πόσο όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο ε, ενεργητικά για άλλους τρόπους, ας πούμε, σύγκριση των των επιδόσεων ή των αποτελεσμάτων ε, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ε, και άλλα σώματα που, το που, προβαίνουν σε αυτές τις ε, διαδικασίες αλλά και άλλοι μηχανισμοί και στο ΝΟΗΕ και στο Συμβούλιο το, της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Θέλετε να κάνετε περώτηση, όχι, ωραία, ευχαριστώ. Ωραία, τώρα να προχωρήσουμε με την κυρία Χόλμαγερ και πάλι. Εσείς θα πάρετε το βραβείο των περισσότερων ερωτήσεων σήμερα. Όχι, εντάξει, τότε ο Τσάμπα Σογκόρ. It's ε, <coughs> agency reports Διαβάζουμε τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, οι αναλύσεις, οι εκθέσεις σε σχέση με τις διακρίσεις, ε, για άτομα που ανήκουν σε παραδοσιακές εθνοτικές μειονότητες. Δεν ξέρω ε, γιατί, γιατί υπάρχουν πολλές διακρίσεις, όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και σε επίπεδο νομοθεσίας. Βλέπετε εσείς κάποια δυνατότητα να ε, κρατήσουν τα κάτι μέλη της υποσχέσεις τους, δηλαδή τα κριτήρια μετά την Κοπενχάγη. Ευχαριστώ, πάντο, όπως πάντα σύντομος. Έχετε δύο λεπτά. Ναι, μια ερώτηση που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή γιατί έχω δουλέψει συγκεκριμένα ε, για τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Όπως ξέρετε, οι εθνικές μειονότητες τώρα πλέον αναφέρονται όχι μόνο στο χάρτη, αλλά και στις προτεραιότητες δράσης, ιδιαίτερα και συγκεκριμένα σε σχέση με τις διακρίσεις ε, ε, και τους νόμους κατά αυτών. Ξέρουμε όμως ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη δευτερογενής νομοθεσία που να είναι και ε, το μεγάλο ερώτημα είναι που με έχει απασχολήσει και εμένα γιατί είμαι και ε, λετωνή και Σουηδή πίκος. είναι κατά πόσο αυτό ισχύει και γιατί τη, ε, ε, κατά πόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνουν και τις μειονότητες και τα δικαιώματα αυτών. Ε, αυτό μπορεί να ισχύει για τα νέα κατημέλια, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο για τα παλαιά, για ιστορικούς λόγους. Πάντως, ε, και βέβαια ε, είχαμε και το ερώτημα που βέβαια στο Κοινοβουλίο και τις εθνικές μειονότητες ε, τη συγκέντρωση των πληροφοριών που υπάρχουν, αλλά και το θέμα του πώς το συγκεκριμένο πολιετές πλαίσιο με όλες τις διαφορετικές ε, πληροφορίες που περιλαμβάνονται εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο τη συλλογή πληροφοριών. Ε, ε, ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από τους σοσιαλιστές, από την κυρία Λόρισταν. Ευχαριστώ πολύ. Συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την προηγούμενη ερώτηση, αλλά δεν αφορά ακριβώς τις μειονότητες, αλλά τους μετανάστες. Ξεκινήσατε ε, με τη μετανάστευση τους, ε, του δεσάσυλου και τα λοιπά. Τι μπορεί να γίνει για την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και τι μπορεί να κάνει οργανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα για να επηρεάσει όλη αυτή την κατάσταση. είναι πίγωνο ο χαρακτήρας του ζητήματος αυτού και το ΦΡΑ ήδη από πέρσι μιλούσε για αυτά τα θέματα στην αιτήσια του διάσκεψη ώστε να πιστήσει την προσοχή, να αυξήσει την ερωτότητα αυτών των θεμάτων και συλλέγοντας στοιχεία ώστε να δείξει που υπάρχουν τα πολύ σοβαρά αυτά προβλήματα στο, για τα συστήματα ασύλου, την εφαρμογή του σχετικής νομοθεσίας αλλά και τους παράνομους μετανάστες και όλα τα σχετικά προβλήματα οι στρατηγικές που υπάρχουν και η ατζέντα για τη μετανάστευση φαίνεται λογικό και ο οργανισμός μας να παίξει κάποιο ρόλο ώστε να δοθεί συνέχεια στα θέματα που περιλαμβάνονται εκεί και αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς που ενεργούν σε αυτό το τομέα δεν θέλουμε να κάνουμε επικάλυψη ή να ε, ε, μπούμε στα χωράφια άλλων. Πάντως ε, μπορεί να γίνει δουλειά και ο οργανισμός μας θα δώσει επιπλέον πληροφορίες, επιπλέον ανάλυση για την κατάσταση που επικρατεί επί τόπου. Να παρακολουθεί δηλαδή τις πληροφορίες αλλά και να τροφοδοτεί με πληροφορίες πιο συστηματικά ώστε να αναπτυχθεί αυτή ε, το μεγάλο θεματολόγιο που θα είναι πιο γενικό και θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα σημαντικά ζητήματα. χωρίς να πιστοδρομήσουμε ε, ε, από προηγούμενους, ορισμούς, ο οργανισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των πληροφοριών που υπάρχουν από τις, από τις πρωτοβουλίες των διαφόρων ε, θεσμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Γιατί καταφέραμε. Εάν δεν είχατε μείνει, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση. Πραγματικά... Ε, μπορούμε και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να συνδυάζουμε τη συζήτηση των σημαντικών θεμάτων την πέμπτη απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους όσους μείνατε λοιπόν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Στις 2 Ιουλίου θα γίνει ψηφοφορία. Κυρία Ολοκληρώθηκε τώρα η ακρόαση και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι.